Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο κομμάτι της εργασίας μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης για τα επόμενα 7 χρόνια, 2014-2020. έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο κάπως έχει ανατραπεί και το πρόγραμμα το οποίο έχει διατυπωθεί ως έρασμος για όλους το έχουμε επηρεάσει προς την κατάλληλη κατεύθυνση. Πάνω από χίλιες τροπολογίες έχουμε. Και αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι δεν μπορέσατε να τροποποιήσετε το δικό μου έγγραφο εργασίας, αλλά περιοριστήκαμε στο να τροποποιούμε το έγγραφο της Κομισιόν. Πολλές τροπολογίες λοιπόν είναι ταυτόσιμες. Τις έχουμε ομαδοποιήσει και έχουμε επίση καταφέρει να καταλήξουμε σε πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Πρόκειται για ένα επταετές πρόγραμμα και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το επεξεργαστούμε εντατικά ώστε να είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το 2014. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης συγητές για την συνεργασία τους. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει παραταξιακό χαρακτήρα. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα για τις επερχόμενες γενναίες. Και όπως καταλάβατε έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες για μένα είναι πιο απλά τα πράγματα, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούτε προσεκτικά, γιατί σε ορισμένα σημεία θα πρέπει να πηδήξω 5 ή 10 σελίδες. Θα χρειαστεί λοιπόν λίγος χρόνος για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα κάνω αργά την ψηφοφορία για να μην χάσουμε τον μπούσουλα. Αν έχετε λοιπόν όλοι τις, τις κάρτες σας μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 263, δική μου τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ, κατά. 236, κατά. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14 έμπλ υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 14 υπέρ κατά άποχες δεκτή 17. υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται Ήτρε 13 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 315 στην επόμενη σελίδα 315-316 είναι μαζί υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 314 και έμπλου 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 314 και έμπλου 16 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτές. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην 18. Ήτρε 18. Υπέρ. Κατά. Α, πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 320. Υπέρ. Ναι, ναι, και εγώ ήμουν υπέρ. Ήμουν υπέρ. Δεν το είχα καταγράψει αυτό. Υπέρ, 320 Κατά αποχές δεκτή. Έμπλ 18 υπέρ κατά αποχές έλχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15-9 γίνεται δεκτή. 19, έμπλ 19, υπέρ, κατά, απόχες απορρίπτεται. 324 υπέρ κατά αποχές άσχητη άσχετη ψηφοφορία πέρας 12-12 απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 325 υπέρ κατά αποχές έλεγχος αυτή την ψηφοφορία. Πέρας. 15-9 γίνεται δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. υπέρ. Κατά. Αποχές. 3.29. υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 326 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 330 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλη 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλη 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 331 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο. αρθει την ψηφοφορία. Πέρας. 13.11 γίνεται δεκτή. Έμπλικος 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.35 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 3.35 πέρας 18.8 ε, δεκτή Εμπλ 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλικος 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλικος 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.37 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε έλεγχο άρχιδη ψηφοφορία πέρας 16-10 γίνεται δεκτή έμπλη 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3.40 <coughs> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί 21 με 25. 21 μέχρι 25 παρακαλώ ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η έμπλη 29 είναι και αυτή η ταυτόσημη 343 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 343 πέρας 16-10 γίνεται δεκτή 26 υπέρ κατά Άλλη μια φορά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 26. Πέρας. 13-12 γίνεται δεκτή. 3.48, επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 345, 346, 347 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτονται 27 και έμπλ 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 350 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 351 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 351. Πέρας. 13-11 γίνεται δεκτή. 29 και 3-52 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεκτές. 3-54 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12-12 απορρίπτεται. Πάλι, πάλι, πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία για την 354. Πέρασε. 13-12 γίνεται δεκτή. Ευχαριστώ Σίλβια. Τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 359 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 έμπλη υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές δεκτή 363 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σύμβαστη 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην ήτρε 20 που είναι στη σελίδα 16 σελίδα 16 Ήτρε 20 Η 16 είναι μετά τη σελίδα 15 λέει η πρόεδρος Σελίδα 16 κάτω, Ήτρε 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ. Κατά. Απόχη. Χαθήκατε, χάσατε. Λοιπόν, πηγαίνετε στη σελίδα 16. Έχετε άλλη αριθμίση. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Εντάξει. Τη βρήκατε? Να ξαναρχίσω. Η 20. Η 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Στην σελίδα 17. Στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πήραμε δύο σελίδες και πάμε στην 390. ...390, μια ή δύο σελίδες αργότερα. Ψήφι υπέρ, κατά. Απόχες δεκτή. 391. Υπέρ κατά αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. 3.91. Ήβο, δεν θα ψηφίσεις. 3.91. Κύριε Μπέκερ, ούτε εσείς. Πέρασε ψηφοφορία 11.15 απορρίπτεται. Ήτρε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 392 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 24. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί 24. Όχι. Ήτρα 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 400, δύο σελίδες πιο πέρα. 400. Φρανθίσκο Χωσέ Μιλάν Μον, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στην Ήτρε 26, δύο σελίδες αργότερα. Ήτρε 26. υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 27, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 413, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2, Αλφόνς Γκρέζ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 28. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κάτω στο τέλος της σελίδας, έμπλ 51. Υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Έμπλ 52. Υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Απόχες δεκτή. Συμβιβαστική 5. Σε δύο σελίδες. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άλλες δύο σελίδες θα πηδήξουμε τώρα. 4.90. Ψήφι υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Αρχίζουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 17.9. Απορρίπτεται. 4.42 στην επόμενη σελίδα. Νεβεντάλοβα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4.51. Επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άλλες δύο σελίδες. 4. Όχι. 478. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 486. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 466. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 467. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 468 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 469 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 470 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 491 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Στην 491 άρχεται. 10,16 10-16 απορρίπτεται. Ή 329 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 492 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΒ11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στην επόμενη σελίδα 493 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μήπως μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία πίσω οι κλητήρες, παρακαλώ. 508. Τέσσερις σελίδες αργότερα. 508. Έμα Μακλάρκιν, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 509, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 5.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλεξτε 1 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 5.10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο για την 510. Άρχεται. Πέρας. 10 με 16 απορρίπτεται. Βλέπω ακόμα, λέει η πρόεδρος. 511 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 514 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεβε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο σελίδες αργότερα στην ΙΤΡΕ 35. Είτε 35, 38, όχι, 35 λέει η πρόεδρος. Εμένα λέει 35 το χαρτί μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 35. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, Ήτρε είναι Επιτροπή Βιομηχανίας και Έμπλη είναι Επιτροπή Απασχόλησης. Βέβαια είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης έχουμε αυτές, τις, αυτά τα ακρόνημα μέσα στο κοινοβούλιο για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. 35 ψηφίσαμε. Προχωρούμε. Ήτρε 38. Μια μισή σελίδα μπροστά. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5.35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται μια σελίδα αργότερα, 547. Υπέρ, κατά, απόχέ. έλεγχος. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. 14-11 απορρίπτεται. 5-49. Εγώ είμαι κατά. Δεν υπάρχει ένδειξη εδώ. Συ, είμαι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 548 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήτρε 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 έμπλ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλ έμπλ όχι 69 εκπίπτει έμπλ 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 138 υπέρ Ναι, ναι, όχι. Ναι, ναι, πάμε στην 72. Έχετε δίκιο. Έμπλε 72, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5.58. 58, υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία στο δεύτερο τμήμα της 558. Πέρας. 17-9 απορρίπτεται. 5-5, συγγνώμη, 5-60 μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 5, δική μου, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Τροπολογία 5 προφορική. Άρχεται η ψηφοφορία. Προφορική τροπολογία 5 της εισηγήτριας. <coughs> ναι, ναι. Πέρασε. Ωραία. Τέμπε 15. Στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12-12 απορρίπτεται. 5-61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5-62. 5-64 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5-63 έχει αποσυρθεί ή 3-42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5-65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 566 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 567 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 568 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 569 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ξέχασαμε κάτι. Συγγνώμη, έχω ξεχάσει την 562 πενεράμπα του υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πού είμαστε τώρα? Έμπλε 74 υπέρ κατά αποχές τεκτή 573 όπως η 143 κτλ. Είναι πολλές ταυτόσιμες τροπολογίες. Όλες συμπούρμπουλε οι τροπολογίες μετά την 573. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 575 και έμπλε 76. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές προφορική, όχι, 1.45, συγγνώμη. 1.45 και 5.76 και ιτρε 46 μαζί. Όλες αυτές οι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 5.70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 572 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 570. Πέρας. 3 με 24. Απορρίπτεται. Μα γιατί, γιατί, γιατί δέχεστε να υποστείτε μια τέτοια ήττα. Δεν το, δεν είπαμε κακή, εν πάση περιπτώσει. 578 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρ. 577 συγγνώμη ήταν αυτό. Υπέρ. Κατά 146 και έμπλε 78 υπέρ. Κατά και η 578 επίσης. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στη συμβιβαστική 10 πολύ μακρύτερα. Τέσσερις σελίδες αργότερα. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 11 τρεις σελίδες αργότερα. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλο 83, τέσσερις, τέσσερις σελίδες αργότερα. Έμπλο 83, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 653, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 178, υπέρ, κατά και η 645 είναι ταυτόσιμη. Α, εκπίπτει. Α, μάλιστα. Πάμε στην 179. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. Ήταν ταυτόσιμη με την 660. 647 Μπεναράμπα του υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πηγαίνουμε τώρα 6 στην 6.48. Α, απορρίφθηκε αυτή. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. 180 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6.48 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 6.58 έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί εν πάση περιπτώσει 6.58. 6.55 υπέρ κατά <clears throat> αποχές έλεγχος για την 655. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκαέξι-δεκά απορρίπτεται. 650 υπέρ, κατά, συγγνώμη, 183 ήταν αυτή. 650 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά απόχες δεκτή. 661 υπέρ κατά απόχες δεκτή. 184, καθώς και 652 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο σελίδες αργότερα 674 674 Liam Aylward υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 675 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 681 έχει αποσυρθεί ωραία όχι Δεν έχει καλυφθεί η προφορική τροποποίηση. Μια, στι... μια στιγμή λέει πρόεδρος. Ναι, ναι, πρέπει να πάμε στη συμβαστική 13 τώρα. αρχίζω να εκνευρίζομαι. Σύμβαστη 13. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6.95 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6.98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο για την 6.98. Υπέρ. Ναι, ναι. Αν πέρασε ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 697. Υπέρ. Κατά. Αποχές. «701 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «702 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τουλάχιστον 4 σελίδες αργότερα στην 86 έμπλ. Το βρήκατε? Πολλές σελίδες, πολλές σελίδες. Πολλές σελίδες αργότερα λέει πρώην. Έμπλο 86. Το βρήκατε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2-0-2. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 17 συγγνώμη. Δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλο 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλε 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλε 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. προφορική τροποποίηση από την Καταρίνα Νεβαντόλεβα ε, για την 764. Ψήφι υπέρ. Δεν υπάρχει στον κατάλογο. Όχι. Μα νόμιζα ότι είχατε μια προφορική τροπολογία. Όχι, δεν υπάρχει. Την έχετε αποσύρει. Η 764 έχει αποσύρθει. 765 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 766 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 υπέρ κατά αποχές δεκτή budget όχι 767 767 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 768 και budget 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 206 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 770 υπέρ κατά έλεγχος για την 770 άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. 17-13 γίνεται δεκτή. Δέλε 18 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία για την ΔΕΒΕ 18. Πέρας. 16-14 δεκτή. 72 772, 773, 74 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 16 σε δύο σελίδες. υπέρ της συμβαστική 16 κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 782 σε δύο σελίδες. Πέτα κάμερα ρεβέρτ. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 783 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 784 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Αρχή την ψηφοφορια πέρασε Πέρας. 13-16 απορρίπτεται. 785, τώρα είμαι υπέρ για το επόμενο. 785, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 787 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14-13 γίνεται δεκτή. Έμπλ 93. Υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές απορρίπτεται. Budget 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 797. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάτσε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 207 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 208 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 798 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 798. 9, 8 πέρας 18, 12 δεκτή συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην 101 έμπλ, στην επόμενη σελίδα. Στο τέλος της επόμενης σελίδας. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.17 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ή 60 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 807 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 808 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. <clears throat> Ή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 809 σε δύο κομμάτια. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές αδεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Θα το ελέγξουμε το δεύτερο κομμάτι της 809. Α, είναι ψηφοφορία. 14 14-15 απορρίπτεται. Έμπλ. Όχι, όχι. Πάμε στην 810. Και την ΤΕΒΕ 21 που ταυτίζονται υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2-19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 811 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 813 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8-14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2-20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 815 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σύμβαση 18 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή πάμε στην 22 ε, 20 όχι πάμε στην 222 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεν το έχετε αυτό το πράγμα. Στην επόμενη σελίδα. Του, του, του. Η 222 δηλαδή. 819 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 820 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 223 υπέρ κατά αποχές δεκτή 821 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Απορρίπτεται. 14 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.25 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχή την ψηφοφορία. Πέρας. 21 με 9 παράξενο. Αυτό γίνεται δεκτή. Budget 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8.23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.26 έχει αποσυρθεί. Υπάρχει εδώ μια προφορική τροπολογία. Μπορείτε να διαβάσετε. Δεν μπορείτε. Ε. Έχει κάποιο την προφορική τροπολογία τη Κατερίνας. Εγώ θα μπορούσα να σας τη διαβάσω. Ακούστε με λοιπόν. Η κατανομή των πιστώσεων για το πρόγραμμα πρέπει να καλύπτει συγκεκριμένες και βιώσιμες ε, επιδοτήσεις σε ευρωπαϊκές οργανώσεις δραστήριες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αυτό το οποίο θέλει είναι να βγάλουμε τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όχι γιατί είμαστε κατά του αθλητισμού, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Ελπίζω λοιπόν να είστε όλοι υπέρ, γιατί εγώ είμαι υπέρ, οπότε πρέπει και εσείς. Λοιπόν, δεκτή. υπέρ, κατά. Από δεκτή. 109 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 8, 27 και 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 8, 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8, 30 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία 8.30 πέρας 8.30 14-14 απορρίπτεται. Ήτρε 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Ήτρε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8-31 υπέρ. Κατά. Κατά. απορριπτεται απορρίπτεται. 8-32 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. Ήτρε 7 υπέρ. Αποχέ Αποχές δεκτή. 2-28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήτε 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 833 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροποποίηση, τροπολογία 8-9 της συζήτησης υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8.34 και 35 και 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 8.37 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Για την 837 έρχεται η ψηφοφορία. 837. περας 10.17 10-17 απορρίπτεται. 841 υπέρ. Κατά απόχες δεκτή. 2. Όχι, όχι. Πάμε στην Ήτρα 1. Πάμε στην Ήτρα 1. Στην επόμενη σελίδα. Ήτρα 1. Πού είναι η τρένα. Η τρένα, να ναι, στην επόμενη σελίδα πράγματι. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. In, when we voted 234, 234 την υπερψηφίσαμε. Και μετά πρέπει να πάμε στην Ήτρε 1. Αλλά δεν αληθεύει αυτό. Δεν πρέπει να πάμε στην Ήτρε 1. Γιατί έχω κάνει ενδιαμέσως μια προφορική τροπολογία. Η τροπολογία 2 στην επόμενη σελίδα. Θα σας τη διαβάσω αν θέλετε. Προηγουμένως όμως έχουμε τροπολογία 241. Κάσλα. Ψήφι υπέρ του 241. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η δική μου προφορική τροπολογία τώρα. Αν θυμάμαι καλά, η ιδέα μου ήταν να κρατήσουμε τη διαβίου εκμάθηση. Μετά είπα να τα αλλάξουμε όμως. Σε αυτή όμως την αιτιολογική σκέψη εξακολουθεί να υπάρχει διαβίου εκμάθηση και δεν αναφέρουμε ε, τα, ε, τα ονόματα των υπολείπων. Οπότε, εξακολουθεί να υπάρχει αιτιολογική σκέψη για τη διαβίου ε, εκμάθηση. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτή την τροπολογική τροπολογία υπέρ. Υπέρ της προφορικής τροπολογίας 2 της κυρίας Πακ. Κατά. Κατά. Αποχές. Κυρία Βριζού, έχετε... Προ... Για ποιο, νούμε, για ποιο αριθμό τροπολογίας μιλάμε. Προφορική τροπολογία 2 μου είπαν εμένα. Ναι, προφορική τροπολογία 2. Ε, τότε είναι του κυρίου Αλφόνση, δεν δική σας. Όχι, πρέπει να δείτε την αιτιολογική σκέψη 3. Λέει, το βλέπετε, 241 την απορρίψαμε. Μετά έχουμε την προφορική τροπολογία 2. Προφορική τροπολογία 2. You did the It's correct here. You see two. Πάμε στην 240. Ναι, τόλβα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήτρε δύο Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Την Ήτρε να την ψηφίσαμε. Εκπίπτει. Α, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. 2.42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. DV1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. EMPL 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. EMPL 3 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.48 και 2.49 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. ΔΒ2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.51 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2.50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.52 υπέρ. Κατά 2.52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.53 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.64 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 264. Πέρας. 17-9 απορρίπτεται. 2.65 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Τρία της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16-11 εγκρίνεται. 2 60, όχι 268, όχι 273, 273 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 273. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14-13 γίνεται δεκτή. 274. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έμπλ 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήτρε 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δε, απορρίπτεται. 276. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 275. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.77 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή δεκτή, 6 υπέρ κατά αποχές δε απορρίπτεται 2.78 υπέρ έλεγχος για την ή 6 ή 6 απερίφθη 2.78 χωρίς μικρόφωνο κυρία Βερζία Δεν σας καταλαβαίνω. Πάω πολύ γρήγορα. Θα το κάνω πιο αργά. Συγγνώμη κύριε Βεζιά. Πού ήμασταν. Ήτρε 6. Να σας τα πω γαλλικά για να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Ήτρε 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν τα λέω γαλλικά. MP6. MP6. Υπέρ. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 280. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλεπτα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τέσσερα της υπέρ κατά αποχές δεκτή. 281 και έμπλοχτο που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές. Δεβετρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 282 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εμπλ, Θέλετε να ελέγξετε τη 282. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία στην 282. Πέρας. Δεκατρία δώδεκα. Μάλιστα. Αλλά είχα δίκιο παρόλα αυτά. Έμπλε νέα υπέρ κατά αποχές το 2.83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία προφορική 13 της εισηγητρίας. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Όχι, όχι. Πάμε στην Ήτρε 7. Οι άλλες εκπίπτουν. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.87 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μα 16-10. Απορρίπτεται. 2-88 υπέρ. Κατά αποχές. 2-93 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2-89 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 2-89. Πέρας. 14-13 γίνεται δεκτή. 2.90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλ 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή τρε 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.92 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.94 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12-15 απορρίπτεται. 2.95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην budget 4 στο τέλος της σελίδας. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 11. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.99 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Budget 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΔΕΒΕ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 303 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλου 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 305 υπέρ κατά αποχές δεκτή 306 υπέρ κατά αποχές δεκτή 307 υπέρ κατά αποχές δεκτή budget 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή budget 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή budget 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 308 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 309 υπέρ κατά απόχες έλεγχος. γιατί την 309 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 1116, 310 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 12 της εισηγήτριας υπέρ κατά απόχες δεκτή και η τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία λέει και στα γαλλικά και στα αγγλικά. Πάμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την τελική ψηφοφορία. Πέρασε. 23 με 1 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Έχουμε, έχουμε ακόμα την... Ε, δεν έχουμε τελειώσει. Το νομοθετικό ψήφισμα η τροπολογία budget 1. Okay. Nur damit Είμαι εναντίον των δύο τροπολογιών του προπολογισμού, την budget 1 και budget 2, δεν το έχω σημειώσει. Budget 1, υπέρ, κατά, υπέρ της budget 1, κατά, μα δεν βλέπω κανένα σηκώνει το χέρι του, υπέρ της budget 1, υπέρ, Κατά. Μα πείτε ότι είστε κατά. Ελάτε, πείτε ότι είστε κατά. Στο τέλος, στο τέλος του καταλόγου. Στο τέλος του καταλόγου έχουμε και τις δύο αυτές τροπολογίες που πρέπει να ψηφίσουμε. Πρέπει να ψηφίσετε. Γιατί έχονται από την Επιτροπή Προϋπολισμών. Άλλη μια φορά υπέρ της ε, budget 1. Κατά αποχές, έλεγχος, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 13-13 απορρίπτονται. Budget 2, υπέρ. Κατά. Έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας με την ίδια πλειοψηφία 13-13 απορρίπτονται. Παρακαλώ. Διαδικαστικό. Θέλω να γραφούν στα πρακτικά ότι η Πρόεδρος τέσσερις φορές έθεσε σε ψηφοφορία την τροπολογία αυτή του προϋπολογισμού. Ήταν τρεις φορές σαφές ότι υπερψηφίστηκε, αλλά στη συνέχεια στην ηλεκτρονική ψηφοφορία έφτασε σε μία ισοψηφία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια μαζική χειραγώγηση της ψηφοφορίας το να θέτετε τέσσερις φορές την ίδια τροπολογία σε ψηφοφορία. Μα δεν πρόκειται αγαπητές συνάδελφοι για κάτι τέτοιο. Ζήτησα να ψηφιστούν ηλεκτρονικά αυτές τις τροπολογίες γιατί δεν ήταν σαφές πώς πηγαίναν οι τροπολογίες και γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν ξέρανε πού βρισκόντουσαν αυτές τις τροπολογίες. Λυπάμαι για την άποψή σας, αλλά δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Κύριε Μπέλετ. Ήθελα απλώ να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε, ότι υπήρχε πολλή σύγχυση. Δεν ήταν σαφέ ε, πού ακριβώ ψηφίζαμε, ε, σε ποια σελίδα είμαστε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πού ακριβώ ήμασταν και τι ψηφίζαμε κάθε φορά. Άλλε δύο Στο τέλο, στο τέλο, στο τέλο. Δυστυχώς δεν είναι σαφές για όλους. Τελική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Υπέρ. Α, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. 21 υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές. Και τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα, ε, αποστροποποιήθηκε στο σύνολό του, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «21 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές». Τέλος. Σας ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Κομισιόν. Είχαμε Είχαμε κάποιες δύσκολες συζητήσεις στην αρχή όταν επεξεργαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Καταφέραμε όμως να καταλήξουμε σε κάποιες ε, λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα τον κύριο Κορέλ και όλους τους συνεργάτες τους. Νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν την ίδια άποψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ήρθε ο κύριος Τάκουλα. Για να δούμε. Σας δίνω το λόγο να μας πείτε ορισμένα πράγματα για την Ευρώπη, για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, Ντόρις, που σήμερα ήρθα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα με τις διαδηλώσεις έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ντόρις για την δουλειά σου για τον έρασμο για όλους. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η δουλειά αυτή. Σας ευχαριστούμε. Δεν θέλω να καθυστερήσω την ψηφοφορία, θέλω όμως να κάνω μερικά σχόλια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, το είπε και η Πρόεδρος, γιατί με βοήθησαν. Θα είναι πραγματικά μια πρόκληση αυτή η έκθεση στο μέλλον και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Με την Επιτροπή και το Συμβούλιο εννοώ. Πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους για να τελειοποιηθεί το πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση. Καταλήξαμε σε μερικούς συμβιβασμούς. Δεν συμφώνησαν όλες οι ομάδες δυστυχώς, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχει ο πολιτικός βίος. Υπήρχαν κάποια ευαίσθητα σημεία Καταλαβαίνω την ε, προφορική τροπολογία η οποία κατατέθηκε σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω γαλλικά, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το τμήμα του πολιτικού διαλόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ του συναδέλφου που συνεργάστηκαν μαζί μου και που απέσυραν κάποιε από τι τροπολογίε του. Να ευχαριστώ και τη γραμματεία. Γιατί βοήθησαν πάρα, βοήθησε πάρα πολύ και δούλεψε και εκείνη πολύ σκληρά. και τον Μάρτιν και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους της γραμματείας, τους συναδέλφους του στη γραμματεία. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω βέβαια και την ομάδα των φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους. Ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτή την έκθεση. Η διαδικασία δεν είναι η συναπόφαση. Ε, ε, καλούμαστε απλώς ε, να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας σε αυτά που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι η διαδικασία θα πρέπει να είναι διαφορετική. Θα μπορούσε να είχε συμμετάσχει το Κοινοβούλιο περισσότερο. Τέλος πάντων δεν συνέβη αυτό. Εμείς θα προσπαθήσουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή. Μας είπε ο εισηγητής ότι δεν καταλαβαίνει γαλλικά. Η Μαρή Κριστίν Βερζιά, ο Λόταρ Μπίσκι και η Νέζ Ζουμπέρ, ε, εκ μέρους της ΓΚΟΕ, υπέβαλαν μια τροπολογία. Διαφωνούν με την έκθεση και αποφάσισαν ε, εν είδη παραρτήματος να υποβάλουν ένα κείμενο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα έγγραφα μειοψηφία. Συμμετείχε η ΓΚΟΕ στις ε, εργασίες για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέει αυτό το κείμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πω ότι από πολιτικής απόψεως η Γκουε είχε ένα πρόβλημα με αυτό το κείμενο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω αν η κυρία Βερζιά θέλει να πάρει το λόγο. Μπορείτε να πάρετε το λόγο αν θέλετε. Ναι. Απλώς για να εξηγήσω τη θέση μας. Καταρχάς, Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη μνήμη της ιστορίας, τέλος πάντων το καθήκον της ε, μνήμης. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει οι πολιτικοί να ξαναγράψουν την ιστορία και όταν οι πολιτικοί ουσιαστικά μιλούν για καθήκον της μνήμης που είναι ένα πραγματικό θέμα, δεν πρέπει να ε, περιορίζουν τα πράγματα, να θέτουν περιορισμούς. Εμείς διαφωνούμε με όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όποια και να είναι. Ε, γνωρίζετε ότι στην ομάδα μας υπάρχουν κάποιοι ε, κομμουνιστές, πρώην κομμουνιστές. Δεν είναι όμως η μόνη. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναγραφεί η ιστορία ε, μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ε, το καθήκον της, ε, της μνήμης δεν είναι μόνο εναντίον των ολοκληρωτικών καθεστώτων, αλλά των ολοκληρωτικών καθεστώτων που υπήρξαν στα εδάφη μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την μνήμη της απεικιοκρατικής ιστορίας, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν αναφέρεται και γι' αυτό υποβάλαμε αυτή την τροπολογία. Εμείς παραμένουμε στην παραδοσιακή ε, άποψη, στην αρχική άποψη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην αρχική πρόταση ε, να μιλούν μόνο για ολοκληρωτικά καθεστώτα και δεν αναφέρονται στο σταλινισμό, στο φασισμό και ούτε συμπεριλαμβάνουν αυτά στον, στα ολοκληρωτικά καθεστώτα υπήρχαν ε, κομμουνιστές, ε, ε, όμως υπήρχαν και κομμουνιστές οι οποίοι με την ζωή τους πλήρωσαν τον αγώνα τους εναντίον του ναζισμού. Δεν γίνεται το ολοκαύτωμα να μπαίνει στην ίδια μοίρα ε, με ε, τον ε, κομμουνισμό. Εγώ νομίζω ότι είναι πραγματικά από ιστορική απόψεως απαράδεκτο και δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι ο κομμουνισμός είναι το ίδιο πράγμα με τον ναζισμό που ήταν μια ιδιαιτερότητα της ιστορίας που είχε ως αποτέλεσμα το ολοκαύτωμα. Τόσοι Εβραίοι χάθηκαν στο ολοκαύτωμα και εμείς ως ΓΟΕ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε συμφωνήσουμε με το κείμενο αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ενδιαφέρουσα θα ήταν αυτή η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να, το την οργανώσουμε για μια μελλοντική συζήτηση. Μας εξηγήσατε τη θέση σας, ε, ε, τη θέση της μειοψηφίας. Μας εξηγήσατε ε, την άποψή σας. Θα δεχθούμε αυτό που μας υποβάλατε. Περάσουμε, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Αύκο 1. Υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αύκο 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159 το ίδιο πράγμα. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12 κατά 10 ε, υπέρ απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές. Budget 6. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 12 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 24 και 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίπε 13 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, 10 κατά, Οι φιλελεύθεροι έχουν μία ψήφο παραπάνω. Όχι. Κύριε Βάτιμο. Εγώ θα ψηφίσω με την αριστερά εδώ. Δεν είμαι εναντίον, απλά αλλάξατε θέση και δεν σας βλέπαμε. Και ψήφιζε κάποιος άλλος στη θέση σας. Ε, 26. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 στην επόμενη σελίδα Αύκο 12 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την ΑΦΚΟ 12. Πέρας. 18-6. Εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, έναρξη ψηφοφορίας για την 176. Πέρας. 22-3. Εγκρίνεται. Αύκο 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικής. Πέραση της ψηφοφορίας. 11-15 απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πρέπει να σηκώνετε καλά τα χεράκια. 20 υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 ή μάλλον λίμπε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 και 31 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 181 και την 31. Πέρας της ψηφοφορίας 17-7 εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας. 19-6 ε, αν σηκώνατε τα χεράκια καλύτερα, δεν θα χρειαζόταν να περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. 183 έχει αποσυρθεί. 197 πάμε τώρα, υπέρ. Κατά αποχές, Απορρίπτεται. Λίμπε 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αύκο 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ Κατά. Α, Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 11. Πέρας. Μάλιστα, εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Δεν δουλεύει το σύστημα. Μήπως να πάτε στη διπλανή θέση. Απορρίπτεται. Λίπε 17 υπέρ κατά 18 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αύκο 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 199 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΛΥΠΕ 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αύκο 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 16-8. Εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, γκρίνεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπη 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας Πέρας. 13-12 εγκρίνεται. 2-14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 243 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρασε. Καφέ παρακαλώ. Merci bien. 13 zu 11 απορρίπτεται. 2.21 υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. Λείπει 24 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. Λείπει 25 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. Λείπει 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 εισηγητής υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2-2-2 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας 16-7 γίνεται δεκτή budget 8 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 2-23 υπέρ 2-23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 μαζί με 2, 24, 25 και 23 κατά αποχές δεκτή και οι άλλες επίσης εγκρίνονται φυσικά. Budget 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Not to be voted. 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή και η 2.32 συμβαστή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.38 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.41. Τι να ελέγξετε, τι θέλετε να ελέγξετε. Τη 2.38. Εντάξει. 2.38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16-9 εγινε δεκτή. 2-41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 52. 52. Πέρας ψηφοφορίας. 14-10 εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 για την 242. Α. Μάλλον δεν περνάμε στη συμβαστική 14 τώρα. Κατά αποχές δεκτή. 27 ΑΦΚΟ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 30. Πώς. Παρακαλώ. Για τη συμβαστική 15. Α, συγγνώμη. Έπρεπε να ψηφίσουμε την 55. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην Λίμπε 30 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίπε 31. Πού να είναι αυτή. Λίπε 31, στο τέλος της σελίδας. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 58. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της 58. Πέρας ψηφοφορίας. 12-19 δεκτή. 2-5-5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2-56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για τη 2-56. Άρχεται η ψηφοφορία. 256. Άρχεται η ψηφοφορία και κλείνει επίση η ψηφοφορία. 13 νέα απορρίπτεται. Η 60 υπέρ κατά απόχέ. έλεγχο για την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. 14 νέα δεκτή. Αύκο 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίπε 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αύκο 30, όχι, όχι, εκπίπτει, εκπίπτει. Α, πάμε στην... Ε, παρακαλώ. 2.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αύκο 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή λίμπε 33 όχι 2.59 όχι εκπίπτει και αυτή λίμπε 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αύκο 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αύκο 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίπε 36 υπέρ κατά αποχές ελ, ελέγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για τη Λίπε 36. Πέρας. Δεκαεπτά δεκτή. 66 με 261, 262 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 68 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Not to be voted. Δεν ψηφίζεται 69. 70 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. εκπίπτουν οι άλλες. 71 ως 77 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Εύκο 35 δεν ψηφίστε. 79 υπέρ κατά απόχες δεκτή. 80 μέχρι 95. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες αυτές μαζί. Όχι. Παρακαλώ. Ε, 85 υπέρ. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίντ. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 92 υπέρ κατά αποχε... εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε από την 80 έως την 95 τις ψηφίζουμε όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Λίμπε 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εν... απορρίπτεται. Λίμπε 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 97 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 97 πέρας απορρίπτεται 98 και αύκο 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 99 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 14-9 εγκρίνονται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την Λίμπε. Άρχεται ψηφοφορία. περα 15 Ναι. απορρίπτεται. Σύμβαστη 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 107. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή αυκό 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 116-115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Λι... 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή Αύκο 5 υπέρ κατά αποχές δεκτές Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 117 Κατά απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 8. Άρχεται η ψηφοφορία. <clears throat> Τέρας της ψηφοφορίας. 15-9 γίνεται δεκτή, 9 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 126 υπέρ. 127 μάλλον, ναι, ξέπεσε 126 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αύκο 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 130 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. 12-12 απορρίπτεται. Αύκο 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Αύκο 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυκο 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή όχι όχι εκπίπτει 132 πάμε στην λίμπε 5 κατά υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη λίμπε 5 16-8 γίνεται δεκτή. Budget 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 135 υπέρ εκπίπτει. Έντεκα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12, 136, 137 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές. 138 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12-12 απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. 17-5 με μία αποχή. Πάμε στο σχέδιο ψηφίσματος. Νομοθετικό ψήφισμα λοιπόν. Έχουμε Budget 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το νομοθετικό ψήφισμα άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. 17-4 με 3 αποχές σας ευχαριστώ. Τα μάλα. Thank you very much, Hanu. Thank you all for making this compromise. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν που καταλήξαμε ε, γρήγορα σχετικά. Θα ήθελε ο κ. Στάκουλα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για την παρανόηση η οποία δημιουργήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει μια παρανόηση αυτό είναι κάτι το οποίο θίγει όλο τον κόσμο. Πάντως η βασική ιδέα πίσω από το πρόγραμμα αυτό είναι η ανάκτηση της ευρωπαϊκής του διάστασης Νομίζω λοιπόν ότι καλά πήγαμε και ε, είναι καλό το ότι πολλές πολιτικές ομάδες το στηρίζουν. Ε, Εμείς λοιπόν καταγράφουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ελπίζουμε ότι και η Κομισιόν θα το πράξει και μαζί με το Συμβούλιο θα συνεχίσει μια τακτική διαδικασία. Όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν, γιατί θα περάσουμε στο σημείο της ημέρησης διάταξης παριθμών 9. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι όσοι θέλουν να κάνουν κατηδίαν συζητήσεις, παρακαλώ να φύγουν. Κυρία Μπεναραμπατού, παρακαλώ να βγείτε έξω από την αίθουσα αν θέλετε να συζητήσετε ιδιωτικά. Καλώς λοιπόν, περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Κουλτούρας για το 2014-2020. 2020-2013, συγγνώμη. Πρόκειται για μια αναβαρχίδα της πολιτικής πολιτισμού το θέμα της πολιτιστικής πρωτεύουσα. Δεν είναι μονάχα το να προβάλλουμε μια πρωτεύουσα, αλλά μέσα από αυτή την πόλη πρέπει να προβληθεί η ευρωπαϊκή κουλτούρα και η διαφορετικότητα και η πολυμορφία των ευρωπαϊκών πολιτιστικών στοιχείων. Είναι σημαντικό να επιληφθούμε αυτού του προγράμματος και να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι μετά το 2019, γιατί μέχρι το 2019 έχουν γίνει οι επιλογές των χωρών όπου θα βρίσκονται οι πολιτιστικές αυτές πρωτεύουσες, το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε επέκεινα του 2013 αν θα έχουμε μία πόλη, δύο πόλεις, πολλές πόλεις ή αν θα χρησιμοποιήσουμε Μία άλλη ιδέα. Είναι σημαντικό λοιπόν να καθορίσουμε καλύτερα τη διαδικασία. Ο κύριος Κουρία έχει κάνει μια πρώτη παρουσίαση και επανέρχεται τώρα. Έχει το λόγο. Και παρακαλώ τους συναδέλφους από τους φιλελεύθερους να σταματήσουν. Μόρτεν, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σιωπή. Εγώ θα προτιμούσα να, φύγει, να μείνεις, αλλά αν θες φύγε. Ο Μάρκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που δεχθήκατε και το αίτημά μου να συζητηθεί η αίτησή μου λίγο νωρίτερα. Γιατί μετά πρέπει να πάω στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών όπου είμαι σκιώδης εισηγητής. Η ανακοίνωση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι μια καλή ανακοίνωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει σαν βάση για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες μικρές βελτιώσεις. Συναντήθηκα με εκπροσώπους της Επιτροπής, τους ευχαριστώ. Ο διάλογος έχει δηλαδή ήδη ξεκινήσει. Για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει πριν από οτιδήποτε άλλο να σχεδιάσουμε το πλαίσιο του συζήτησης αυτής και να δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα έτσι ώστε να αναζητήσουμε τους μελλοντικούς προσανατολισμούς. Μέχρι τώρα και με κάποιες μικρές εξαιρέσεις θα έλεγα, οι πόλεις οι οποίες έχουν γίνει ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολιτισμού είχαν θα έλεγα πολλές επισκέψεις επισκεπτών αλλά δυστυχώς τον χρόνο που ακολουθεί την χρονιά της ανάληψης ε, της ε, ιδιότητας αυτής, ε, δυστυχώς οι αριθμοί επανέρχονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια διαχρονική θα έλεγα ωφέλεια. Ενώ οι χώρες, οι πόλεις που φιλοξενούν τους Ολυμπιακούς τουλάχιστον για 7 χρόνια ε, ε, προκαλούν θα έλεγα επισκέψεις ε, επισκεπτών μάλλον στις συγκεκριμένες πόλεις ενώ τώρα στην περίπτωσή μας δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα το 1 τρίτο των πόλεων που πήραν τον τίτλο αυτό οικονομικά έχουν χάσει χρήματα, δεν έχουν κερδίσει το 1 τρίτο έχουν έρθει στα ίσια τους εισαγωγικά και μόνο το 1 τρίτο επίσης μπόρεσαν μέσω της ανάπτυξης υποδομών να έχουν ένα σχετικό οικονομικό κέρδος για την πόλη. Σε ποιες περιπτώσεις λοιπόν οι εμπειρίες αυτές της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας του Πολιτισμού πήγανε ε, θα έλεγα πολύ καλά. Αυτό συμβαίνει όταν σε επίπεδο οργάνωσης, προγραμματισμού υπάρχει συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντισμός κτλ. Και αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο, πολύ συνοπτικά βέβαια, της κατάστασης μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης δύο στοιχεία κριτικής απέναντι σε αυτά τα οποία έχω. Καταρχά Καταρχάς, η περίοδος. Εμείς συζητάμε σήμερα μία πρόταση η οποία θα ισχύσει μέχρι το 2033. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πόσο η δουλειά την οποία κάνουμε σήμερα και την οποία θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου είναι κάτι το τόσο καλό που θα ισχύσει για 20 χρόνια. Όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα γνωρίζουμε ότι έχουν διάρκεια 7 ετή και το πρόγραμμα τώρα του, της πολιτιστικής πρωτεύουσας μέχρι το 2033 μου φαίνεται σαν στόχος κάπως υπερβολικά φιλόδοξος Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε μια ενδιάμεση χρονική περίοδο και κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αυτής χρονικής στιγμής, όχι μόνο μέσω μιας απλής ανακοίνωσης της Επιτροπής αλλά και του Κοινοβουλίου, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Γιατί εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, δημοσιονομικές εγγυήσεις για το τι θα συμβεί μέχρι το 2033. Εμείς μέχρι τώρα ε, προχωράμε μέσω ακριβώς της απονομής θα έλεγα ενός βραβείου 1,5 εκατομμύριο σε κάθε πόλη αλλά τη απουσία ενός πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ήδη για τα επόμενα 7 χρόνια είναι δύσκολα τα πράγματα. Μέχρι τώρα το, 1900, το 2033 είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και εδώ θα ήθελα τις απόψεις των συναδέλφων για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν αυτό είναι πρόβλημα μόνο για μένα ή και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν από κοινού να το αντιμετωπίσουμε. Τι θα μου άρεσε να προσθέσω εγώ στην ανακοίνωση την οποία έχει ήδη κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, θα ήθελα να αναφερθώ στην όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Είπαμε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την επιτυχία του θεσμού. Ε, θα προτιμούσα η Ευρωπαϊκή Διάσταση, και αυτό το υπογραμμίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η Ευρωπαϊκή Διάσταση να τονιστεί ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα η πόλη η οποία θα επιλεγεί να είναι μια ε, θα έλεγα επιλογή η οποία να σέβεται τις οδηγίες της κοινοτικές, τις ρυθμίσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας, τις οδηγίες για το περιβάλλον, της ανακύκλωσης των αποβλήτων. Θα έλεγα, θα ήθελα να είναι μια πολύ καλή καγαθή, θα έλεγα, πρότυπο και σε όλα αυτά τα επίπεδα. Αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση να περιλαμβάνει θα έλεγα και παραδείγματα πόλεων που έχουν ήδη διαμορφώσει επαφές τα προηγούμενα χρόνια με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, να μην γίνονται όλα την τελευταία στιγμή δηλαδή από μία πόλη, αλλά να ανήκει η πόλη αυτή σε ένα δίκτυο επαφών με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι ώστε να διευκολύνει θα έλεγα τις επαφές της με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες και να μην ξεκινά τις επαφές την στιγμή αυτή. Κάποιες πόλεις έχουν καταθέσει ίσως καλά προγράμματα και πήραν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας, αλλά πολύ συχνά η δυνατότητα υποδοχής των επισκεπτών δεν ήταν στο κατάλληλο επίπεδο και διαμορφώθηκαν αρκετά προβλήματα και μερικές φορές και κάποιες αντιθέσεις ανάμεσα στους πολίτες και τους επισκέπτες. Γιατί όπως είπα ακριβώς δεν υπήρχε η δυνατότητα μιας σωστής μορφής οργάνωσης. Θα ήταν λοιπόν καλό οι πόλεις να δείξουν ότι έχουν μια δυνατότητα μακροημέρευσης αυτών των προγραμμάτων τους να μην λειτουργεί αποκλειστικά μόνο το σύστημα αυτό υποδοχής για ένα χρόνο που ισχύει ο τίτλος της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας. Θα ήθελα επίσης τη στιγμή που θα κατατεθεί η υποψηφιότητα να υπάρξει ε, σύμφωνη γνώμη του πολιτικού πανοράματος ε, της διακυβέρνησης της πόλης. Πολλές φορές βλέπουμε ότι τη στιγμή που καταθέτει την πρόταση ο Δήμος μιας πόλης και τη στιγμή κατά την οποία γίνεται η πόλη αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, ε, αυτός που κατέθεσε την αίτηση είναι στην αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια υποψηφιότητα η οποία να συνυπογράφεται από όλο το φάσμα της ε, διοικητικής πολιτικής σκηνής της πόλης. Έχουμε μπροστά μας ε, και μία χρηματοδότηση σχετικά περιορισμένη, 1,5 εκατομμύριο, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί το ποσό αυτό και θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χώρα, η, οποία, η πόλη η οποία θα αναγνωριστεί σαν πρωτεύουσα πολιτιστική να έχει δυνατότητα καλύτερης και αμεσότερης πρόσβασης στα διαφθρωτικά ταμεία και σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο περιφερειακό. Όταν ζητά δηλαδή χρηματοδοτήσεις να υπάρχει κατά προτεραιότητα δυνατότητα να πάρει αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να εντάξουμε ε, επίσης ε, και το θέμα της επιστημονικής έρευνας στη διάσταση της πολιτιστικής πρωτεύουσας, γιατί η έρευνα και ο πολιτισμός πηγαίνουν από κοινού. Ε, να μπορεί δηλαδή να κάνει τις αιτήσει ε, που απαιτούνται μια πόλη υποψηφία όταν ε, η, η έρευνα που γίνεται η επιστημονική στη συγκεκριμένη πόλη έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Αναφέρθηκα πολύ συνοπτικά λοιπόν σε μια πρώτη, σε μια πρώτη περιγραφή του θέματος, είναι και η πρώτη συζήτηση που θα γίνει, θα ακούσω με προσοχή τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Απλά ένα μικρό κατάλογο θα έλεγα θεμάτων σας έθεσα με στόχο τη βελτίωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επαναλαμβάνω όμως είναι μια καλή πρόταση και είναι μια σωστή βάση για τον διάλογο που ξεκινήσαμε ήδη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλήξουμε σε μια θα έλεγα συνενετική θέση. Ευχαριστώ Μάρκο. Η κυρία Καμ... Ε, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι καλά νέα το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την πολιτική της πολιτιστικής πρωτεύουσα. Χαίρομαι γιατί συμμετείχα σε πολλές αντιπροσωπείες που επισκέφθηκαν αυτές τις πρωτεύουσε, τις πολιτιστικές και αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά ότι υπάρχει μία προστιθέμενη αξία και αποτελεσματικότητα. Εδώ και 25 χρόνια βέβαια ε, έχουμε δει τα πλεονεκτήματα αλλά και τα όρια αυτής, ε, αυτού του θεσμού. Τρία βασικά στοιχεία. Καταρχάς υπάρχει ένα πρόβλημα δημοσιονομικό στο πλαίσιο μιας Ευρώπης ε, που περνάει η κρίση, υπάρχει το θέμα της τουριστικής προώθησης που υπερέχει των υπολείπων πτυχών και υπάρχει επίσης και μια διαφορά μεταξύ αυτού που υπόσχονται οι πόλεις και αυτού που τελικά ε, κάνουν. Νομίζω ότι ο εισηγητής ε, ανέφερε κάποιες ε, διόδους που πρέπει να σκεφτούμε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει, πολιτιστη... υπάρχει προστιθέμενη αξία για την πολιτιστική πρωτεύουσα και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν Εγώ είμαι μέλος και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και βλέπουμε ότι για την αστική ανάπτυξη θα μπορούσε η πολιτιστική πρωτεύουσα να είναι ε, μια σημαντική ε, διαδικασία. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία για την ε, αναδιάρθρωση των άστεων και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη γιατί είναι και ένα στοιχείο διάρκειας. Επίσης ε, μπορεί να είναι αυτά τα αποτελέσματα ε, λόγω του ότι μία πόλη έχει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, μπορεί να γίνουν σημαντικές αλλαγές, μπορεί να προσελκύσει τουριστική ε, πολύ τουριστική κίνηση και υπάρχουν και λιγότερο απτές πτυχές, όπως είναι για παράδειγμα η βελτίωση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών πολιτιστικών φορέων. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ και όπως είπε και ο Μάρκο, η ευρωπαϊκή διάσταση δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ εμφανής. Βλέπουμε περισσότερο την πολιτιστική διάσταση, ε, την τουριστική πτυχή, τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες προβάλλει η πόλη και ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε τα κριτήρια που μπορούν να ευνοήσουν την επιτυχία και τη διάρκεια. Τι μπορεί να προτείνει η Ευρώπη ώστε ε, να υπάρξουν μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα ωφέλη. Υπάρχει το δημοσιονομικό πρόβλημα. Ε, να δούμε για παράδειγμα τον προπολογισμό της Μασαλίας του 2013 ε, είναι πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο που έχουμε εμείς είναι πραγματικά ψίχουλα και δεν νομίζω ότι ε, θα μπορέσουμε να, θα, μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε όλα αυτά που θέλουμε και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, ε μόχλευσης που θέλουμε να έχουμε. Ενδεχομένως ε, να μπορούμε να επικαλεστούμε τη συμπληρωματικότητα με τις πολιτικές ε, υπόλοιπε υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για παράδειγμα τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως ε, τα πολιτιστικά κονδύλια Μήπως θα έπρεπε να έχουμε μία πολιτιστική μόνο πρωτεύουσα κάθε χρόνο και, κάθε χρόνο και όλα τα κονδύλια να πηγαίνουν σε μία και όχι σε δύο πόλεις. Είναι ένα ζήτημα προπολογισμού, το ξαναείπα. Ευχαριστώ. Η Πέτρα. Η Πέτρα, ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον Μάρκο για τις προτάσεις του να ζητήσω συγγνώμη για τον Ήβαν, ο οποίο δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα, είναι ο σκιώδη συζητητή μα. Μου έχει δώσει ορισμένε ε, σημειώσεις, λέει ότι θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό. Να διατηρηθεί λοιπόν αυτός ο χρονολογικός κατάλογος τον οποίο έχει προτείνει η Κομισιόν Θα ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία αλλιώς αν έχουμε τελείως ανοιχτό κατάλογο. Και η Καταλήνα έχει χαιρετήσει τα νέα διατυπωμένα κριτήρια της Κομισιόν γιατί με τον τρόπο αυτό θα είναι σαφέστερο για τις ε, πόλεις και τις περιοχές που είναι υποψήφιες ποιες απαιτήσει θα πρέπει να ικανοποιήσουν και τι πρέπει να εξασφαλίσουν και τι κατεύθυνση θα πρέπει να έχουν Όλα αυτά λοιπόν είναι ιδιαίτερα θετικά και εγώ συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι το θέμα της ε, ανάπτυξης των πόλεων με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και μια μεγαλύτερη ε, συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Ο Μπάρκο ήδη ανέφερε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον προϋπολογισμό Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι για ένα δήμο, για μια πόλη να οργανώσει ένα τέτοιο έτος πολιτιστικής πρωτεύουσας χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά υπάρχει πάντα και η υποστήριξη του κράτους μέλους. <clears throat> Θα ήθελα από τη δική μου πλευρά να κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αποδεκτό η Κομισιόν να είναι αυτή η οποία θα αναλάβει την ευθύνη της επιλογής των πολιτιστικών πρωτευουσών και έτσι θα πάρει αυτή την αρμοδιότητα από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε σε όλες τις περιπτώσεις να εξετάσουμε και τις πολιτιστικές πολιτικές της κάθε χώρας και της κάθε περιφέρειας και να εξασφαλίσουμε ότι είναι υπεύθυνε και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει και μία διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όπως υπήρξε στο παρελθόν. Και φυσικά <clears throat> η πολιτική πολιτισμού είναι μία πολιτική που υπόκειται στην επικουρικότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 167 της Συνθήκης της ε, Λισαβόνας και είναι σαφές ότι οι αρμοδιότητες παραμένουν στα κράτη-μέλη και αυτό σημαίνει ότι και οικονομικά, χρηματοδοτικά θα πρέπει να παίξουν ρόλο τα κράτη-μέλη. Και επίσης δεν είμαι σίγουρη για τα κριτήρια τα οποία προτείνει η Κομισιόν για την Ελλανόδικο Επιτροπή. Κάτι άλλο το οποίο είναι σαφές από την εμπειρία που έχουμε στο παρελθόν είναι το εξής. Η Κομισιόν να μην είναι μονάχα η πολιτιστική πρωτεύουσα, η πόλη η ίδια, αλλά και η περιραίουσα περιοχή. Για μένα όμως αυτή η έννοια είναι κάπως ασαφής. Θα προτιμούσα να μιλάμε για μια περιφέρεια. Άμα σκεφτούμε το 2010, που δεν ήταν μόνο πόλεις και οι περιφέρειές τους, οι περιοχές γύρω τους, αλλά ήταν περιφέρειες που είχαν βραδευτεί, νομίζω ότι θα πρέπει και στο μέλλον να υπάρχει δυνατότητα οι πολιτιστικές περιφέρειες της Ευρώπης να είναι υποψήφιες και όχι μονάχα αστικοί σχηματισμοί, ακόμα και διαμεθοριακές περιφέρειες να μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο αυτό. Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι εφικτό, γιατί είναι κάτι το οποίο ευθυγραμμίζεται ιδιαίτερα με την ευρωπαϊστική σκέψη και μένα νομίζω ότι για μένα μου φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε και στις περιφέρειες την εμπειρία αυτή και όπως έγινε και με την περιοχή του Σάρλουξ. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ θετικά και θα πρέπει να θεσπίσουμε λοιπόν σαφή κριτήρια. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Εγώ γνωρίζω τα θέματα αυτά από δική μου προσωπική πείρα. Λέει ότι, λέει ο Μάρκο, ότι μόνο το 1 τρίτο αυτών των πόλεων έχει δώσει κάποια συνέχεια και έχει εκμεταλλευτεί το καθεστώς αυτό. Για να γίνει όμως αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει κοινωνική συμπερίληψη, ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις, να φτιάξουμε πολιτιστικά έργα κτλ. Αλλά αυτά οδηγούν σε δημιουργία χρέους και αυτό δεν έχει νόημα. Χρειάζεται να χρειάστηκε χρόνο ώστε το Κοινοβούλιο να κατανοήσει, όπω κατανοήσαμε στη δεκαετία του 90 μαζί με την Κομισιόν, ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια νέα κατεύθυνση, να δώσουμε ε, έμφαση στην ε, βιωσιμότητα και την αηφορία, την κοινωνική συμπερίληψη και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε ένα πρόβλημα. 1,5 εκατομμύρια έχουμε μονάχα. Είναι μία σταγόν εν το ωκεανό ή εν τη ερήμο. Αυτά δεν επαρκούν φυσικά για μια τέτοια διοργάνωση, η οποία είναι διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα εκπροσωπεί μια περιφέρεια, εκπροσωπεί ένα κράτος. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος να δείξει το ενδιαφέρον του, ώστε η χώρα αυτή, η πόλη συγγνώμη αυτή, να αποτελέσει και τη βιτρίνα του σύνολου κράτους. Δεν μπορεί βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά. Κάτι ακόμα. Αυτό που είπε ο Μάρκο μέχρι το 2033. Είναι σαφές. Είχαμε ήδη ξεκινήσει το 2000 και τώρα έχουμε 27 και του χρόνου 28 κράτη. Αν λοιπόν θέλουμε η κάθε χώρα να συμμετάσχει, χρειαζόμαστε 28 χρόνια, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από το 2033. Και είχε αποφασιστεί ότι θα έχουμε μία μορφή προγραμματισμού για 15 χρόνια και δεν θα γίνεται με ένα αυθαίρετο τρόπο, αλλά δεν έχουν τότε, όταν είχε αποφασιστεί αυτό για τα 15 χρόνια, δεν είχαν έρθει ακόμα οι 10 νέε χώρε, οι 12 νέε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε πει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτιστική πρωτεύουσα από το, τη Δυτική Ευρώπη και μια από την Ανατολική Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε αν θα πρέπει να συνεχίσουμε με δύο πολιτιστικέ πρωτεύουσε ή αν θα πρέπει να υπάρχουν άλλε δυνατότητε, τρει, ξέρω εγώ. Ή αν υπάρχει μια δυνατότητα για περιφέρειες, για διαμεθοριακή υποψηφιότητα. Αν έχουμε μια περιοχή, ε, μια περιφέρεια που έχει μια πόλη στην πρώτη χώρα, μια στη δεύτερη χώρα, μια στη τρίτη χώρα, τότε μπορούμε με τον τρόπο αυτό να υποστηρίξουμε τρεις πόλεις με σε εισαγωγικά σε ένα χρόνο. Υπάρχει λοιπόν πολύ υλικό για σκέψη και αναστοχασμό για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα μια τέτοια διοργάνωση. Αυτό λοιπόν το οποίο είχαμε κάνει στο τέλος δεκαετίας του 80 να έχουμε ένα πολιτιστικό μήνα θα ήταν πολύ χρήσιμο γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε και σε άλλους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν περισσότερο. Άκουσα πολύ καλά αυτά που είπε η Μαρή Τερέζα η οποία ασχολείται με τα διαφορετικά ταμεία. Είναι σημαντικό το θέμα των, ε, της αηφορίας και της κοινωνικής συμπερίληψης, να προωθήσουμε και την απασχολησιμότητα. Δεν είναι λοιπόν θέμα μονάχα πολιτισμού, όσο η απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα. Θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας λοιπόν αυτό και θα πρέπει να πούμε και στις εθνικές κυβερνήσεις ότι δεν πρόκειται μονάχα να περιοριστούν για να διεκδικήσουν το 1,5 εκατομμύριο, αλλά όταν έχουν και άλλα προγράμματα και σχέδια τα οποία αναπτύσσουν, μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσει και από τα διαφορετικά ταμεία. Είναι πολλά λοιπόν αυτά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει όμως να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία γιατί του χρόνου πρέπει να καθορίσουμε τον κατάλογο αυτό. Τα κράτη χρειάζονται τουλάχιστον 4-5 χρόνια χρόνο για να προετοιμάσουν μια πολιτιστική πρωτεύουσα. Πρέπει να τους δώσουμε χρόνο να προετοιμαστούν και γι' αυτό πρέπει να βιαστούμε λιγάκι με την πρότασή μας. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει μια διαδικασία α, διαβούλευσης. Δεν ξέρω τι ακριβώς ε, έχει προκύψει. δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αυτοί με τους οποίους εγώ μίλησα και οι οποίοι έλαβαν μέρος στην διαβούλευση. Αυτό μπορεί να είναι η προφορική τους άποψη, αλλά θα ήθελα να ξέρω εδώ ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για τη διαβούλευση και γενικά για το πρόγραμμα αυτό. Αυτό είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ούτως ή άλλως. Αν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα θετικά που είπατε για τη συνέχεια του προγράμματος και τα θετικά για την πρότασή μας. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή στην πρότασή μας και μετά να σχολιάσω συγκεκριμένα θέματα που έχουν ήδη τεθεί. Καταρχάς, μπορεί να, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η πρότασή μας βασίζεται σε έρευνα, σε διαβούλευση η οποία έγινε επιγραμμικά Είχαμε επίσης και μία διάσκεψη, θα έλεγα, για τα 25 χρόνια του προγράμματος. Υπήρξαν και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, τις οποίες χρησιμοποίησαμε και επίσης χρησιμοποίησαμε επίσης και την εμπειρία μας, γιατί εμείς είμαστε η μνήμη όλων των διαδικασιών επιλογής για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς χρησιμοποιήσαμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και προσπαθήσαμε να καταλήξουμε ε, σε κάποια συμπεράσματα και επί τη βάση, όπως είπα, της διαβούλευσης της δημόσιας η οποία έγινε. Ο λόγος που κάνουμε την πρόταση αυτή τώρα φαίνεται λίγο νωρίς, αλλά το κάνουμε για να επιβεβαιώσουμε, να διασφαλίσουμε ε, την συνέχεια μετά το 2020 γιατί το παρόν πρόγραμμα ε, λύγει το 19. Ε, θα πρέπει έξι χρόνια πριν να ξεκινήσει ο διαγωνισμός όπως ξέρετε οπότε ήδη δηλαδή θα πρέπει να λειτουργήσουν οι νέες διαδικασίες επιλογής από το 2014 με τους νέους τρόπους. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τα στοιχεία που έχουν πάει καλά Έχουμε αρκετή εμπειρία τώρα για πολλά χρόνια και προσπαθούμε να κάνουμε όμως και βελτιώσεις στους τομείς τους οποίους θα μπορούσαμε ε, να είμαστε πιο αποδοτικοί. Ο τίτλος προσδίδει θα έλεγα η ιδιαίτερο πρεστής της πόλης, αλλά αυτό δεν είναι φυσικά κάτι του αυτόματο. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε στην πρότασή μας. Αυτό που θα επιθυμούσαμε είναι κάθε πόλη, πρωτεύουσα του πολιτισμού, να αφήνει τη δική της κληρονομιά επιτυχίας. Κάθε πόλη που συμμετέχει στη διαδικασία, είτε κερδίζει είτε όχι, να κερδίζει κάτι σε, στρατηγική, σε στρατηγικό επίπεδο. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες συμμετέχουν λοιπόν στις διαδικασίες αυτές και γι' αυτό θα πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα θα έλεγε έτσι ώστε να μπορέσουν κάτι να βγάλουν από τη διαδικασία ακόμα και αν δεν επιλογούν. Πέντε συγκεκριμένα θέματα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε στην πρότασή μας. Πρώτον, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επιπλέον κίνητρα για την διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας ανάμεσα στην εποχή που κατατίθεται η πρόταση και τη χρονιά που παίρνει τον τίτλο η πόλη, γιατί ε, έξι χρόνια μεσολαβούν, τέσσερα χρόνια αυτή τη στιγμή πάρει τον τίτλο η πόλη, υπάρχουν φυσικά εκλογές ανάμεσα και εμείς θα θέλαμε να υπάρχει κοινή αποδοχή των προτάσεων αυτών και σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο προϋπολογισμού. Αυτό είναι το πρώτο που θέλουμε, να πετύχουμε τη συνέχεια δηλαδή. Δεύτερον, η κληρονομιά αυτής της ε, προσπάθειας είναι κάτι που εξαρτάται από το μακροπρόθεσμο της στρατηγικής της. Τρίτον, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση, κάτι το οποίο δεν ήταν πάντα δεδομένο. Πολλές φορές κυριαρχούσαν τα τοπικά συμφέροντα. Εμείς επιμένουμε ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα και όχι για μια εθνική πολιτιστική πρωτεύουσα. Ενισχύουμε τις διαδικασίες αξιολόγησης ε, για να υπάρχουν κοινέ θα έλεγα διαδικασίες. Ε, δεν είναι υποχρεωτική αξιολόγηση για τις ίδιες τις πόλεις. Προσπαθούμε να το επιβάλλουμε αυτό, να κάνουμε τις πόλεις να σκέπτονται στρατηγικά και να βλέπουν ε, με ποιους τρόπους τα πλεονεκτήματα τα οποία προσδίδονται στις συγκεκριμένες πόλεις που επιλέγονται να συνεχίζουν και μετά την λήξη ε, της ε, αρχικής περίοδου. Η διαδικασία, όπως είπα, λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια. Θέλουμε εμείς ε, να διατηρήσουμε την ποιότητα την οποία είχαμε μέχρι τώρα. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αλλά απαιτείται να ισχύουν κριτήρια τα οποία θα διασφαλίζουν την ποιότητα αυτή για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα που τέθηκαν από σας Καταρχάς, εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, η γενικότερη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες. Αυτό είναι κάτι που εντάσσουμε στην πρότασή μας. Λεπτομερείς προτάσεις και κριτήρια για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και στην κατάθεση της υποψηφιότητας και στη λειτουργία και επίσης εμπλοκή του πολιτιστικού τομέα της πόλης στις διαδικασίες. Αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε να υπάρχει ένα αίσθημα ιδιοκτησίας ε, των πολιτών ε, στα πλαίσια αυτής της ε, λειτουργίας θα έλεγα και του θεσμού. Έχουμε επίσης συγκεκριμένα κριτήρια και για την εμβέλεια στην οποία, την, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες αυτές διαδικασίες. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί, δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι μειονότητες σαν παράδειγμα. Όλο, όσο και περισσότεροι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν. Τώρα για τη διάρκεια 33% και το 2033 συγγνώμη, ε, εμείς έτσι και αλλιώ θα κάνουμε αξιολογήσεις ανεξάρτητες, ζητάμε να γίνονται, αναπενταετία και θα συμβουλευόμεθα επίσης και την Επιτροπή των Περιφερειών γύρω από αυτές τις αξιολογήσεις. Τώρα για το αν οι πόλεις ε, έχουν τις υποδομές που απαιτούνται, εμείς έχουμε συμπεριλάβει κάποια κριτήρια για την ικανότητά τους αυτή. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιλέγουμε μια πόλη επί τη βάση της διάστασης του πληθυσμού, του μεγέθους του πληθυσμού της. Απ' την άλλη η πόλη θα πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να φιλοξενήσει ένα τέτοιο συμβάν για ένα ολόκληρο χρόνο. Τώρα, για την αηφορία τη χρονική αυτής της ε, λειτουργίας ε, την οποία προωθούμε. Κοιτάξτε, εμείς προωθούμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν θέλω τώρα να εκθέσω λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει σαν παράδειγμα μια υποχρέωση για την πόλη ήδη τη στιγμή της κατάθεσης ε, της υποψηφιότητας να υπάρχει μια πλήρης μακροπρόθεσμη πολιτιστική στρατηγική. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ακόμα και αν η πόλη δεν κερδίσει τον τίτλο, αν μη τι άλλο θα έχουμε επηρεάσει εμείς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτιστική της ανάπτυξη. Τώρα για τις χρηματοδοτήσεις. Έγιναν αρκετά σχόλια για το ύψος των διαφεσίμων ποσών, τα οποία δεν είναι πολύ μεγάλα. Να μην ξεχνάμε ότι στην ουσία παίρνουν έναν τίτλο. Ο τίτλος αυτός αποδίδει οικονομικά. Είναι θα έλεγα κάρτα de visite για πάρα πολλά μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. 1,5 εκατομμύριο είναι αρκετά υψηλό ποσό. Πολύ σωστό ε, είναι ότι κάποιες πόλεις παίρνουν πολλά χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία, 100 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια. Εμείς προσκαλούμε τις πόλεις αυτές να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα και από το Ταμείο Συνοχής. Νομίζω ότι οι πόλεις βλέπουν ότι τα ωφέλη είναι μεγαλύτερα από το κόστος και βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις και οικονομικά κάτι τέτοιο είναι θα έλεγα ιδιαίτερα αποδοτικό. Τώρα, ε, γιατί εμείς ε, ζητάμε να υπάρχει ε, θα έλεγα ε, θέση αποφασιστική της Επιτροπής στη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι του Συμβουλίου. Εμείς έτσι αναγυγνώσκουμε τη συνθήκη ε, της Λισαβόνας. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνουμε εμείς. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένα προηγούμενο με την ετικέτα, την πολιτιστική θα έλεγα, ε, που βασίζεται σε μια επιλογή που γίνεται με, με, πολιτιστικέ πολιτιστικές αξιολογήσεις υπάρχει ένα νομικό θέμα εδώ, αλλά κυρίως υπάρχει ένα πρακτικό θέμα. Επιλέγοντας ε, τη συγκεκριμένη οδό, εμείς παρακολουθούμε την διαδικασία ε, από πολύ κοντά. Ε, οκτώ μήνες μεσολαβούν από τη στιγμή που το πάνελ επιλογής παίρνει την απόφασή του μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης ε, όλη αυτή τη διάρκεια του χρόνου οι πόλεις πρέπει να συνεχίζουν να αυτοαποκαλούνται υποψήφιες πόλεις και ξέρω ότι μερικές φορές υπάρχουν θέματα στον τομέα της χρηματοδότησης γιατί οι πόλεις αγωνιούν για να διασφαλίσουν περισσότερο πιστώσεις. Τώρα, για το κατά πόσον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία ε, της περιφέρειας. Η νομική βάση προβλέπει πόλη, όχι περιφέρεια. Μπορεί όμως να λειτουργήσει στα πλαίσια της περιφέρειας. Εμείς ε, δεν αποκλείουμε την περιφερειακή διάσταση όπως είχε γίνει στο παρελθόν με την ε, κοιλάδα του Ρουρ. Ε, δεν ενδιαφέρονται όλες οι πόλεις να αυτοτοποθετηθούν σε μια περιφέρεια και να οριστούν μέσω αυτής. Πάντως είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα όμως να σας ε, ρωτήσω το εξής. Όπως έχει δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο, εσείς λέτε ποια χώρα, σε ποια χρονιά θα έχει την πολιτιστική πρωτεύουσα. Αυτό αποφασίζεται από το Συμβούλιο. Και η Κομισιόν έχει συμφωνήσει με αυτό από το 2002. Είχε αποφασίσει το Συμβούλιο Ποιε θα είναι οι χώρες μέχρι το 2019 που θα έχουν αυτή την πολιτιστική πρωτεύουσα. Αυτό με την διακριτική του εξουσία, το έχει αποφασίσει το Συμβούλιο και έτσι θα παραμείνει. Αν κατάλαβα καλά, αναφέρεστε στον κατάλογο της γεωγραφικής ε, εναλλαγής είναι παράρτημα στην πρότασή μας, ε, στην οποία, την οποία, στην οποία θα καταλήξουν οι συνομοθέτες, εσείς και το Συμβούλιο. Τρεις αρχές ε, υπήρχαν, αλλά ούτως ή άλλως ο νομοθέτης θα αποφασίσει κατά πόσο θα ακολουθήσει αυτή τη σειρά ή κάποια άλλη. Σας απαντώ στην ερώτησή σας με αυτά που είπα. Κατάλαβα καλά. Δεν είναι θέμα περιεχομένου, λέει η πρόεδρος Πακ όχι για την πόλη, αλλά για το πότε η κάθε χώρα θα, πότε κάθε χώρα θα αναλάβει. Αν είναι ένα θέμα το θα, για το οποίο θα μπορεί να επανέλθει το Κοινοβούλιο, αν εμπίπτει στην απόφαση ή αν είναι το Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει τη χρονολογική σειρά των κρατών που θα ορίσουν την πολιτιστική πρωτεύουσα για να αποφασιστεί η σειρά, η χρονολογική ε, των ε, χωρών. Είναι η δική μας η πρόταση, την οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ο νομοθέτης. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δηλαδή πρέπει να επιβεβαιώσει τη δική μας πρόταση. Μπορείτε βέβαια να κάνετε αλλαγέ, αλλά κάθε κράτος μέλος θα οργανώνει το δικό του εθνικό διαγωνισμό. Μάλιστα, κατάλαβα. Μα δεν το κάναμε έτσι ως τώρα. Μέχρι τώρα το Συμβούλιο αποφάσιζε. Ο κατάλογος των χωρών ο αριθμός, της, ο, τρόπος εναλλαγής τους βασίζεται στη νομική βάση. Αυτό είχαμε αποφασίσει τότε. Αυτό είχαν αποφασίσει οι νομοθέτες τότε. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, προσπαθώ ακόμα να το καταλάβω αυτό. Το θέμα των περιφερειών. Ξέρετε ότι η Κομισιόν η δική μας Επιτροπή δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη όταν το Λουξεμβούργο, μια μικρή χώρα, είχε αναλάβει την ε, πρωτεύουσα, αλλά λέγοντας ότι θέλουμε να έχουμε και άλλες περιοχές μαζί μας. Παραδείγματο χάρη τον Ζάρλαντ στη Γερμανία, την Ρινανία Παλατινάτο, το Βέλγιο ή την περιοχή του Μοζέλ στη Γαλλία. Δεν το θέλανε, αυτό έγινε Κατά τη δική μου άποψη, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε σκέψεις. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την ενδοχώρα μιας περιοχής. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες ξεπερνάνε τα εθνικά σύνορα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν παραγωγικά χάρη τρεις χώρες να συμμετέχουν στην πολιτιστική, διοργάνωση αυτής της πολιτιστικής πρωτεύουσα. Αλλιώς είναι δύσκολο. Αν μια χώρα έχει αναλάβει ήδη το 2012 ε, μια τέτοια πρωτοβουλία και αλλιώς θα μπορέσει μόνο μετά από πέντε χρόνια να το κάνει. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο. Ίσως θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, παραδείγματος χάρη το Άχεν και το Μάστριχ που είναι πολύ κοντά, αν το Μάστριχ γινόταν πολιτιστική πρωτεύουσα και θα ήθελε να πάρει μαζί του και το Άχεν, τότε και πάλι καλύπτεται η Γερμανία και οι κατοχώρες καλύπτονται και πάλι. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα το οποίο να είναι πιο εύκαμπτο από αυτό που έχουμε σήμερα, δηλαδή να πούμε αυτή η χώρα εκείνη τη χρονιά, η άλλη χώρα εκείνη τη χρονιά, θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ευκαμψία. Ιάν. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι το τρέχον σύστημα είναι μάλλον ευέλικτο. Ε, αυτό που θέλουμε είναι μία πόλη να πρωτοστατεί. Από εκεί και πέρα όμως ε, είναι ευέλικτο το σύστημα. Δεν θέλουμε δηλαδή η περιφέρεια να έχει την ε, κυριότητα γιατί τότε θα ήταν ε, άνισος ο διαγωνισμός και δεν θα υπήρχαν διαγωνισμοί σε όλες τις χώρες. Πάντως το Λουξεμβούργο δεν το σταμάτησε κανένας να αποτελεί τμήμα της ευρύτερης περιφέρειας αν όμως θέλετε, αν, όμως, αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι θέλουμε μία πόλη να πρωτοστατεί και αυτό να είναι σαφές. Μπορεί βέβαια αν θέλουν να συμπεριλάβουν ε, τοπικές ε, αρχές πόλης από την ευρύτερη περιοχή. Μία πόλη όμως δεν θέλουμε να έχουμε τέρους σε διάφορες χώρες ε, για την πόλη αυτή, γιατί ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολη η διαχείριση έτσι. Δηλαδή θέλουμε η διαχείριση να γίνεται σε μία συγκεκριμένη πόλη, ώστε να μην είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Πάντως το σύστημα όσο έχει αυτή τη στιγμή είναι μάλλον ευέλικτο. Η Πέτρα κάτι για τις περιφέρειες ακόμα. Νομίζω ότι η επιχειρηματολογία είναι μία η οποία επιβεβαιώνεται από την ε, εμπειρία που είχαμε το 2010. Είχαμε μια τέτοια κατάσταση που είχαμε την εμπλοκή περιφερειών. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε μια περιφέρεια με την έννοια διοικητική μονάδας, μια θεσμοποιημένη μονάδα. Ο στόχος είναι ότι αν αποφασίσουν οι Δήμοι από κοινού να συνεργαστούν με πόλεις ή κοινότητες που βρίσκονται κοντά να μπορούν να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αυτού του είδους. Το 2010 υπήρχαν συνεργασίες 15, 15 πόλεων που λειτουργήσαν πολύ καλά. Οπότε αυτό είναι κάτι ευρύτερο από μία πόλη και την, μαζί με την ενδοχώρα της. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ευελιξία και να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν από μόνα τους τα διοικητικά προβλήματα και να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Αυτό, επομένως, βοηθάει και τη συνεργασία των διαφόρων πόλεων που βρίσκονται σε μια ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω την Κομισιόν να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία και ιδίω, όπως το έχω ξαναπεί, για διαμεθοριακές περιοχές. Μας είπε, παραδείγματος το παράδειγμα η κυρία Πακ του Άχεν και του Μάστριτ, που μπορούν να συνεργαστούν συγχρόνως για να είναι πολιτιστικές πρωτεύουσε. Και έτσι λοιπόν μπορούν όλες οι εμπλεκόμενες πόλεις να έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν και μία προστιθέμενη αξία μέσα εισαγωγικά από τη διοργάνωση αυτή της πολιτιστικής πρωτεύουσα. Επομένως είναι απαραίτητη η περαιτέρω ευελιξία και ευκταία κατά την άποψή μου. Ναι, ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να πω, το 2012 ο τίτλος απονεμήθηκε στο... στην περιοχή Essen-Ruhr. Ε, υπήρχε όμως η δυνατότητα οι υπόλοιπες, οι υπόλοιπες πόλεις να ε, αποτελέσουν τμήμα της ευρύτερης περιφέρειας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ζωηρή συζήτηση. Φαντάζεστε πώς θα πάνε τα πράγματα όταν θα αρχίσουμε, όταν θα σχεδιάσουμε το πρόγραμμα. Μάρκο. Κάποια μικρά σχόλια. Στη χώρα μου σαν παράδειγμα που καταθέτει την υποψηφιότητα για το 19 υπάρχουν πόλεις υποψήφιες οι οποίες φυσικά και εμπλέκουν θα έλεγα την περιφερειακή διάσταση, την περιοχή στην οποία βρίσκονται, εντάσσονται. Και αυτό δημιουργεί ένα δίκτυο το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για την συγκεκριμένη πόλη αλλά και για το σύνολο της περιφέρειας. Η ιδέα αυτή λοιπόν και για τις διαμεθοριακές τέτοιου είδους συνεργασίες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Να δούμε όμως πώς θα το μορφοποιήσουμε. Πάντως όπως είπα έχουμε ξεκινήσει μόλις τώρα. Εγώ θα μείνω σε επαφή και με τους σκιώδεις των υπολείπων πολιτικών ομάδων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική πρόταση μετά από αυτό που άκουσα σήμερα το πρωί. Ωραία, σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Θα παρακολουθήσουμε τα θέματα αυτά. Εγώ ένιωσα κάποια ανακούφιση γιατί μπορούμε να ξέρουμε ότι θα υπάρχει λιγότερη χρηματοδότηση, αλλά μπορούμε να το επεξεργαστούμε καλύτερα το θέμα αυτό. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Ερχόμαστε στο σημείο 8. Αγαπητή Σίλβια, έχω ένα προβληματάκι. Μόνο η κυρία Τρίπελ είναι παρούσα και ο κύριος Μπίσχη από τους σκιώδεις εισηγητές. Ξέρω ότι έχει κάνει τρεις συναντήσεις με τους ε, σκιώδεις εισηγητές δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για 700 τόσες τροπολογίες. Ίσως, αν θες, μπορείς να πεις κάτι για τα θέματα αυτά, γιατί σήμερα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα απουσία των συναδέλφων και ξέρω ότι θες να κάνεις μια εντατική συζήτηση με τους συναδέλφους σε πιο κλειστό κύκλο. Αν θες λοιπόν να κάνεις κάποιες παρουσιάσεις των σημείων όπου υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Παρακαλώ. Λυπάμαι που δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι εδώ, αν και κάποιοι σκιώδη σημαντικοί είναι παρόντες και εκπρόσωποι της Επιτροπής. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία των 477 τροπολογιών, 78. Αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά με αφορμή αυτή τη συζήτηση να ακούσω από τους σκιώδεις και από την Επιτροπή κάποιες διευκρινήσεις ε, γύρω από τις τοπολογίες που θεωρούν ότι είναι οι πιο σημαντικές για αυτούς. Και να έχουμε την δυνατότητα λοιπόν ε, υπό το φως των μελλοντικών συναντήσεων να καταλήξουμε κάπου. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Έχουμε και τις νομοδοτήσεις ε, των Επιτροπών Προϋπολογισμού, Εξωτερικού Εμπορίου και Γυναικών Υπάρχουν πολλές τροπολογίες γιατί αφορούν και το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τη δική μου έκθεση, στην οποία έτσι κι αλλιώς ε, υπάρχουν κάποιες αλλαγές και κάποιες διευκρινήσεις. Νομίζω ότι οι τροπολογίες αυτές μπορούν, ε, θα έλεγα, να αντιμετωπιστούν με μια κάποια ευκολία. Για να μην καθυστερήσουμε άλλο, θα ήθελα να πω ότι οι τροπολογίες ορισμένων τουλάχιστον συναδέλφων επιβεβαιούν την επιθυμία τους να καταστήσουμε πιο συγκεκριμένο και πιο ορατό και πιο ορατά μάλλον τα δύο αυτά προγράμματα. Θα έλεγα ότι οι τροπολογίες ανήκουν σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει σαν στόχο τον εμπλουτισμό μπαίνουν ίσως και σε υπερβολικές λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει διευκρινίζεται σε επίπεδο λεπτομέρειας το κείμενο και ενισχύεται θα έλεγα, εντάσσοντας πιο συγκεκριμένους στόχους και κάποιους πιο συγκεκριμένους ορισμούς και μέτρα. Αναφέρομαι εδώ στους συναδέλφους του ΕΛΚΑ, των φιλελευθέρων, σε αυτά που είπε η κυρία Τρούπελ κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι τροπολογίες, όπως πάρα πολύ συχνά συμβαίνει, επαναλαμβάνονται ή επαναλαμβάνουν πράγματα που καθιστούν, θα έλεγα, το κείμενο πάρα πολύ ε, δυσκίνητο και βαρύ. Ε, θα ήθελα βέβαια οι ιδέες των συναδέλφων να είναι παρούσες, όπως ο διπολιτισμικός διάλογος, κάτι το οποίο απασχολεί πολλούς συναδέλφους, μια καλύτερη διευκρίνηση της φύσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα, τον δημιουργικό και του πολιτισμού. Το λέω και προς τον συνάδελφο Μπίσκι ότι ορισμένοι συνάδελφοι θα έλεγα ε, στην ουσία αναφέρονται κατά αποκλειστικότητα σε θέματα πολιτισμού. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κάποια ε, μορφή ισορροπίας που επιτρέπει και τις ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις του πολιτισμικού τομέα να συμμετέχουν. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι τονίζουν υπερβολικά την προτεραιότητα που έχει ο ραδιοτηλεοπτικός τομέας. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει, θα έλεγα, μια ισορροπία ανάμεσα στον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης. Και φυσικά Υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, ομάδες τροπολογιών, όπως αυτή την οποία υπογραμμίζει η κυρία Τρούπελ, για την αξία που έχει η πολιτιστική κληρονομιά και ο πολιτισμός που θα πρέπει να ισορροπούν με τις προτεραιότητες που έχουμε στον τομέα τον οικονομικό και της ανταγωνιστικότητας. Εγώ προσωπικά θα αξιολογήσω λοιπόν όλες αυτές τις προτάσεις και για τους λεγόμενους πολιτισμικούς πρέσβεις, όπως επίσης και σε κάποιες ε, προσπάθειες και πρωτοβουλίες στον τομέα της ε, κληρονομιάς, όχι της πολιτιστικής, αλλά της ραδιοτηλεοπτικής. Τα λέω όλα αυτά γιατί τελικά θέλω να πω ότι υπάρχει μια ομάδα τροπολογιών η οποία μπορεί να γίνει γενικότερα εύκολα δεκτή. Μια δεύτερη τέτοια ομάδα, εκεί ότι υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες από πλευράς μου να τις δεχτώ γιατί εξασθενούν την έκθεση, εξασθενούν τον ρόλο του Κοινοβουλίου, ε, τροπολογίες που μειώνουν τον προϋπολογισμό, που ε, είναι εναντίον των κατεξουσιοδότηση πράξεων, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ τίθεται το θέμα και των ε, εκθέσεων σε ετήσια βάση. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει και μία τρίτη ομάδα που διευρύνει υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, όπως ο καθορισμός του πλαισίου θα έλεγα, λειτουργίας του προγράμματος, και αυτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για αυτά τα πλαίσια ε, προτείνονται ε, δύο επιπλέον τομείς και από την κυρία Τρούπελ και από τον κύριο Μπίσκι και από την κυρία Παλιαδέλη επίσης ε, να εμπλακεί πλήρως δηλαδή το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πρόγραμμα, κάνοντας διακρίσεις βέβαια στις αρμοδιότητες ε, οι οποίες ανήκουν στα διαφορετικά ταμεία, αλλά παρόλα αυτά ε, δικαιωματικά η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει στο πρόγραμμα αυτό και σε επίπεδο άειλων και σε επίπεδο υλικών αγαθών. Πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε σε θέματα όπως ε, η ιστορική, γαστρονομική διάσταση ε, και σε κάποιους άλλους τομείς και δραστηριότητες όπως οι τουριστικές δραστηριότητες και τα κτλ. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν ανήκουν στον κόσμο της, ε, τον, τον δημιουργικό ε, και στον κόσμο τον πολιτισμικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες προτάσεις, ε, ποικίλε προτάσεις για, το, για τη διεύρυνση του πλαισίου εφαρμογής της πρότασής μας. Εν πάση περιπτώσει εγώ κάνω μια πρόταση την οποία θεωρώ ισόρροπη, αλλά είμαι διατεθειμένη να συζητήσω την πιθανή διεύρυνση του πλαισίου αναφοράς της. Τώρα, Αυτά ήταν τα βασικά, θα έλεγα, χαρακτηριστικά των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλές μπορεί να γίνουν δεκτές και ο κύριος Καβαντά έχει εμβαθύνει στα θέματα αυτά και έχει διακρίνει τα πεδία, ε, τα διαφορετικά των τροπολογιών και σε σχέση με τα ισχύοντα προγράμματα και για τον πολιτισμό και για το ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Άλλοι συνάδελφοι που δεν είναι παρόντες αυτή τη στιγμή προσπάθησαν κατά κάποιο τρόπο να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους τομείς και τις λεγόμενες εγκάρσιες μορφές παραγωγής πολιτισμού ορίζοντας ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Και υπάρχει τώρα και ένα τμήμα των τροπολογιών το οποίο νομίζω είναι εκτός νομικής βάσεως του κανονισμού Αναφέρομαι στο θέμα της ψηφιοποίησης σαν παράδειγμα. Κοιτάξτε, ό,τι ανήκει στις αρμοδιότητες, είτε της Ευρωπαίνα, είτε ε, των διαφορετικών ταμείων, είτε του Ταμείου Συνοχής. Αυτά τα λέγαμε χθε και με την κυρία Νέλη Κρούς. Προφανώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί περισσότερο το θέμα της ψηφιοποίησης, αλλά δεν θα γίνει εδώ αυτό. Εμείς προσπαθούμε να προτείνουμε κάποιες πλατφόρμες στα πλαίσια των οποίων θα προωθήσουμε την καινοτομία περισσότερο. Ε, κάτι άλλο το οποίο είναι εκτός νομικής βάσης είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, τα θέματα των θεωρήσεων εισόδου για καλλιτέχνες από άλλες χώρες και άλλα θέματα που αφορούν άλλα προγράμματα Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά πάρα πολύ σύντομα και γρήγορα γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που ορίζονται στις τροπολογίες εκτός νομικής βάσης. Τώρα βλέπω ότι έχουμε εδώ εκπροσώπους της Επιτροπής και θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει η δυνατότητα περαιτέρω ζήμωσης. Η πρώτη ερώτηση. Εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από τις συναντήσεις τις οποίες είχαμε στα πλαίσια της Επιτροπής Πολιτισμού να κατανοήσει τους λόγους που οδηγούν σε ένα πρόγραμμα πλαίσιο που ισορροπεί από τη μία την καινοτομία των λεγόμενων εγκαρσίων τομέων με μια διεπιστημονική αντιμετώπιση του θέματος, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας πλήρως και συγκεκριμένα κάποια προγράμματα που αφορούν τον πολιτισμό. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα επίπεδο ικανοποιητικό διαλόγου και συνεννόησης με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Για το θέμα τώρα το οικονομικό, στο οποίο έχει θέσει και ο κ. Καβαντά. Νομίζω ότι μετά από την πρόσκληση την οποία πήφθηνε η Πρόεδρος την προηγούμενη φορά, εμείς είχαμε μια χρήσιμη συζήτηση με τους Σκιώδης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφερθήκαμε και στο οικονομικό μέσο, ε, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Καβαντά και τους άλλους συναδέλφους και έχουμε μια βάση για την οποία μπορούμε, με την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαθεσιμότητά της. Μπορούμε να εμβαθύνουμε στον τομέα αυτό της χρηματοδότησης, να καταστήσουμε τη χρηματοδότηση αυτή πιο κατάλληλη ε, για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας που θα ωφελήσει και τις μικρομεσαίες αλλά και τις μικρές πολιτιστικές επιχειρήσεις και να δούμε ακριβώς και τι είδους δάνεια μπορούν να γίνουν ε, αντικείμενο εγγυήσεων. Ένα τελευταίο σημείο αφορά ένα άλλο θέμα το οποίο έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου μετά από κάποιους ανεπίσημους ελέγχους και συζητήσεις που είχα, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με όλους τους συμμετέχοντες στον τομέα αυτό. Είναι ένας τομέας στον οποίο δεν ακούστηκαν πολλά από συναδέλφους, αλλά θα ήθελα να το θέσω. Όλοι επιθυμούμε, όπως και στο πρόγραμμα Erasmus να διευρύνουμε τη συμμετοχή προγραμμάτων όπως το Μέντια, πολιτισμού κτλ προς χώρες ε, τις οποίες θα έλεγα είναι χώρες γειτονίας ή τρίτες χώρες γενικότερα. Είχα κάνει λοιπόν μια πρόταση, να υπάρξει δηλαδή ότι η προϋπόθεση για να συμμετέχει κανείς στο πρόγραμμα Media είναι να επικυρώσει κατά κάποιο τρόπο ή μάλλον όχι να επικυρώσει, να αποδεχθεί την ισχύ των οδηγιών του 2010 για το ραδιοτηλεοπτικό ε, προϊόν, για τη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή και για την τηλεόραση χωρίς σύνορα. Νομίζω ε, ότι λίγες είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Η Ελβετία χρειάστηκε πέντε χρόνια για να μπορέσει να πάρει μέρος και γι' αυτό προτείνω ένα σταδιακό χαρακτήρα εμπλοκής και συμμετοχής των τρίτων χωρών να συμμετέχουν δηλαδή οι χώρες αυτές ακόμα και αν βρίσκονται σε μια προκαταρκτική φάση. So che tema delicato. Volevo solo chiarire e sentire θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έχει τεθεί το θέμα και από δική της πλευρά. Ένα τελευταίο θέμα θα ήθελα να είναι ε, μια προσεκτική αντιμετώπιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπάρχει μια δυσκολία να κατανοήσει κανείς και το θέτουν αυτό πολλοί συνάδελφοι το θέμα της κοινωνικής διάστασης, της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσθέσουμε στα μέτρα τα οποία προτείνουμε, αλλά είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι θα έλεγα των χαρακτηριστικών μιας δημιουργικής και πολιτισμικής Ευρώπης. Συμφωνώ με τους συναδέλφους λοιπόν να βρούμε τρόπο έτσι ώστε να μην ξεπεράσουμε τις αρμοδιότητες μας στον συγκεκριμένο τομέα, να μην επιβαρύνουμε την πρόταση, αλλά να μην αγνοήσουμε το θέμα αυτό της κοινωνικής πολιτιστικής διάστασης. Νομίζω ότι ε, κατά τα άλλα θα συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το θέμα αυτό είναι σημαντικό και βαθιά πολιτικό. Ευχαριστώ, Ντόρις. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Θα ήθελα να σταθώ τώρα πολιτικά σε τρία σημεία, τα οποία για μένα είναι πολύ σημαντικά. Όταν μιλάμε για το νέο αυτό πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, μαζί με το πρόγραμμα για τον πολιτισμό και το πρόγραμμα για τα μέσα, τα οπτικοακουστικά μέσα, εγώ θέλω να κάνω σαφές μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρωπαϊκή 2020, 20 ποιες είναι οι σχέσεις με την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κλάδο και το πολιτιστικό κλάδο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει σε βάρος των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων πολιτιστικού χαρακτήρα. Υπάρχει το πλαίσιο της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας και πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενταχθούν και όλα τα προγράμματά μας για την πολιτιστική πολυμορφία. Θα πρέπει να είναι σαφές λοιπόν ότι δεν θα κάνουμε τίποτα το οποίο θα έρθει σε αντίφαση με το πλαίσιο της UNESCO για την πολιτιστική πρωτοβουλία και κατέστησε και τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα δεύτερο θέμα για την διευκόλυνση χρηματοδότησης. Αν λειτουργήσουν αυτά σωστά, μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και μικρά σχέδια, τα οποία πάντα είχαν δυσκολία να βρουν κεφάλαιο κινδύνου. Αλλά για να μπορέσει αυτό να γίνει αποτελεσματικά, θα πρέπει οι προποθέσει να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια και θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχεται κάποιο, παραδείγματο χάρη, σύμβουλο μια τράπεζα που θέλει να βγάλει ένα ευρώ παραπάνω και ο οποίο δεν θα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα θέματα της κουλτούρας και του πολιτισμού. Θα πρέπει ο τρόπος αυτός που θα γίνει χρηματοδότηση να υποστηρίζει πραγματικά τα μέσα ε, και τη δημιουργία σε πολιτιστικό επίπεδο. Δεν θέλω να είμαι συντηρητική, δεν θέλω να εμποδίσω μια τέτοια κατεύθυνση ένα τέτοιο εγχείρημα. Απλώ θέλω να υπάρχουν οι απαράγραπτε προποθέσει ώστε πράγματι να χρηματοδοτούνται προγράμματα τα οποία έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο και δεν θα πρέπει να αποτρέπει αυτούς οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Τρίτον, έχω καταθέσει και τροπολογίες που προβλέπουν <clears throat> να υπάρξει και μια υποστήριξη στο πρόγραμμα Media και των ε, ε, προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τις ταινίε για παιδιά, με τα πολιτιστικά ε, προγράμματα για παιδιά. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί ιδιαίτερα. <clears throat> Ευχαριστώ. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για τα φιλμ που απευθύνονται σε παιδιά και είχα ξεχάσει να το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, ξέρουμε εμείς σε, σε τι αναφερόμαστε. Ο κύριος Τσβέρ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό. Εγώ όμως θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες και τις φιλοδοξίες της συναδέλφου Κώστα. Επίσης, συμφωνώ και με την τάση απλοποίησης που υπάρχει, κάτι το οποίο σημαίνει μείωση της γραφειοκρατίας και για τους καλλιτέχνες αλλά και για τους οργανωτές. Αιτιολογική σκέψη 23. Αναφέρεται στην απλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και νομίζω ότι η τροπολογία μου ενισχύει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια. Να εξηγηθώ. Μιλάω για τη χρωματοδότηση μέσω ε, καταποκοπήν ποσών. Για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης, τα ποσά αυτά δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ενώ στα, στα πολιτιστικά προγράμματα Υπάρχουν τα ζητήματα μετάφρασης, υπάρχουν πολλές ε, ε, ε και ο λόγος είναι ένα προς τρία. Και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να αμβλυνθούν αυτές οι διαφορές ώστε και να τροποποιηθεί το ε, πρόγραμμα σωστά προς αυτή την κατεύθυνση. Και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει πράγματι να εξασφαλίσουμε ότι όχι μονάχα η δυνατότητα απασχόλησης θα πρέπει να ληφθεί από τα προγράμματα αυτά, αλλά θα πρέπει να έχουμε προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες στον πολιτιστικό τομέα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει πάντα η Κομισιόν. Έχουμε λίγα λεφτά στον τομέα αυτό και είναι πολύ πιο εύκολο να δοθούν αυτά τα λεφτά σε μεγάλα σχέδια. Αυτό είναι πιο εύκολο σε διαχειριστικό επίπεδο. Υπάρχουν ξέρω πολλούς οι οποίοι δεν διεκδικούν πλέον χρηματοδότηση γιατί το χαρτοβασίλειο που πρέπει να συμπληρώσουν είναι τόσο μεγάλο που δεν αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει τα χρήματα τα οποία θα πάρουν. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα για αυτό το πρόγραμμα, ιδίως αν θέλει να υποστηρίξει μικρά α, σχέδια και προγράμματα, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να περιοριστεί η γραφειοκρατία στην οποία υπόκεινται τα προγράμματα αυτά γιατί έτσι χάνουμε και την θετική θέληση των καλλιτεχνών και των δημιουργικών ανθρώπων. Μας ενδιαφέρουν μονάχα τα έγγραφα και οι διατυπώσεις. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να το κατανοήσει ότι η διαδικασία αυτή της διαβούλευσης θα πρέπει να λειτουργήσει κάπως καλύτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βελτιώσει τα πράγματα. Είναι σημαντικό για μας λοιπόν όσο δυνατόν πιο σύντομο να είναι το ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει κανείς ώστε να μην αποτρέπει αυτούς οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αυτές και όχι όλα αυτά να γίνονται προς όφελος των εταιριών consulting. Θα πρέπει να είμαστε φιλικοί προς το χρήστη και φιλικοί προς την κουλτούρα. Και επίσης το σχέδιο αυτό είναι ανοιχτό και για τις χώρες ε, που είναι υποψήφιες για ένταξη. Έχουμε την Ελβετία η οποία παραδοσιακά δεν θέλει να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω ότι μπορεί να υποφελθεί από αυτό το πλαίσιο. Η Κροατία σαν χώρα που έχει προσχωρήσει είναι επίσης επιλέξιμη για αυτά τα σχέδια <coughs> και ξέρω ότι και η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει ζητήσει μέσα στα πλαίσια της γειτονία να ε, επωφεληθεί. Δεν είναι φυσικά υποψήφια ακόμα, αλλά βρίσκεται στο προενταξιακό στάδιο και έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από αυτά τα προγράμματα. Θα είναι χρησιμό λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και φαντάζομαι ότι η κυρία ε, δεν θέλει η Κομισιόν να λάβει το λόγο. Θέλετε, η κυρία Ντασίλβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερη και να επικεντρωθώ στα ερωτήματα που ετέθησαν. Ακούσαμε, διαβάσαμε τις τροπολογίες με πολύ ενδιαφέρον. Μερικές από αυτές εμπλουτίζουν την συζήτηση. Έχουμε κάποια γενικά σχόλια όμως και ειδικότερα να πούμε ότι πολλές από τις τροπολογίες αυτές ε, έχουν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος, κάτι το οποίο πραγματικά ε, θα ήταν ε, σχεδόν αδύνατο να συμβεί χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού και επειδή υπάρχει και επικάλυψη με κάποια άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά και τους τομείς δράσης και θα ήθελα να αναφερθώ στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να διέπεται από αυτό το πρόγραμμα ε, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή. Ορισμένα ζητήματα είναι εντελώς εκτός πεδίο εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα νομοθεσία για τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αδειοδότηση. Ε, το ίδιο θα ίσχυε και για τους στόχους δεν ε, ε, θα μπορούσαμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματο να ασχοληθούμε με ζητήματα Ευρωπαϊκή ηθαγένεια, α πούμε, γιατί υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο εφαρμογή ε, του προγράμματο αυτού, που επικεντρώνεται σε, ένα, σε μια χρηματοδότηση ε, δημιουργίας. Δεν, δεν υποκαθιστά τι πολιτικέ για, για τον πολιτισμό και του σχετικού τομεί που αποτελούν αντικείμενο άλλων εγγράφων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με την πολύ χρήσιμη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμω, ο ορισμό που έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι στενότερος ε, από αυτόν της πράσινη βίβλου και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να διευρυνθεί γιατί υπάρχει ο κίνδυνο να μην μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Το ίδιο θα ισχύει και για τους υποψήφιους δικαιούχους και για κάποια ε, μέτρα ε, στο πλαίσιο του προγράμματος. Όσον αφορά το θέμα που έθεσε η κυρία Κώστα και ε, το γενικότερο θέμα που αφορά τους στόχους, σημειώνουμε ότι κάποιες από τις τροπολογίες προτείνουν ε, διέρεση σε δύο υποπρογράμματα. Εμείς δεν συμφωνούμε. Πιστεύουμε ότι η πρόταση είναι εξισορροπημένη, δεν θέτει να αμφιβόλο την εγγενή, την εγγενή αξία του πολιτισμού και λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές αξίες, ε, ε, την κοινωνική, ε, την πολιτιστική καταλαβαίνουμε βέβαια τις διαφορές ε, μεταξύ ε, των του, οπτικοακουστικού τομέα και των άλλων δημιουργικών τομέων, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται πλήρως ε, στα προγράμματα και στους δείκτες που ασχολούνται ειδικά με αυτούς τους τομείς. Όλοι οι τομείς έχουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες προκλήσεις, κατακαιρματισμός της αγοράς, ε, τάση ψηφιοποίησης, ε, δυσκολία πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά κονδύλια και έχουν παρόμοιους στόχους. Ο τρίτος πυλώνας μπορεί να δίνει κάποιες δυνατότητες διατομεικών ε, προσπαθειών όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη πολύ συντονισμένης εργασίας ε, για ε, την υποστήριξη ε, των δεδομένων, όπως επίσης και την χορήγηση εγγύησεων. Πιστεύουμε ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι ένα αποτέλεσμα και των τριών αυτών στοιχείων έχουμε τους στόχους μας ε, και έχουμε και την υποχρέωση ε, κάποιων δικτών, ούτως ή άλλως ήδη, το να προσθέσουμε περισσότερους θα δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που θα επέλυε. Όσον αφορά την ευθυγράμμιση τώρα των γραφείων υποστήριξης, ε, αυτές, αυτοί, αυτές οι τρεις, ε, αυτές, αυτή η τριπλή προσέγγιση που ε, προτείνουμε δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα ενιαίο σημείο επαφή χωρί την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, Απλώ θα είναι καλύτερη ευαισθητοποίηση σε όλους τους πολιτιστικού και δημιουργικού τομεί και θα υπάρξει και εξοικονόμηση όσον αφορά τα ε, γραφεία υποστήριξης. Επίσης δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στις περιφέρειες και στα κράτη-μέλη να έχουν ε, μια παρουσία ε, δικαιούχων σε τοπικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και η ε, δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων. Ένα ακόμη θέμα που αφορά την πολιτιστική πτυχή ο τρόπος ε, με τον οποίο έχει οριστεί η ε, χρηματοδότηση, το επίπεδο χρηματοδότησης είναι διαφορετικός ε, από την αρχική διάκριση μεταξύ ετήσιου και πολιετούς χαρακτήρα του προπολογισμού και ακόμη και στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων είναι διετής η πρόβλεψη των κονδυλίων γιατί η ετήσιος χαρακτήρας είναι πάρα πολύ περιοριστικός. για τα οπτικοακουστικά ζητήματα, ε, για τα οπτικοακουστικά, τα ζητήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας ε, εξετάζονται ε, και το πέμπτο πρόγραμμα που αφορά ειδικότερα την παραγωγή δεν θεωρείται ότι πρέπει να σύμπεριληφθεί. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή, καλό είναι να δούμε τους δείκτες ε, που έχουν προταθεί και επανερχόμενοι στους στόχους, οι περισσότεροι δείκτες ε, θα ήταν προβληματικοί. Ο αριθμός των δικτών ε, που εισάγονται δεν θα ήταν μετρήσιμοι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα παραβιάζουμε την νομική βάση και δεν θα μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ε, δείκτες αυτούς. Το θέμα των εφαρμοστικών πράξεων επίσης είναι γνωστό και θα έλεγα απλώς ότι η μόνη εφαρμοστική ε, πράξη είναι αυτή που προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος ε, του ετησίου και όσον αφορά την διευκόλυνση εγγυήσεων, το επίπεδο λεπτομέρειας που προτείνεται σε πολλές από τις τροπολογίες θα δημιουργούσε προβλήματα. Πιστεύουμε επίσης ότι δεν θα πρέπει να αναφερθόμαστε σε συγκεκριμένους ε, φορείς όπως η UNIC και η UFSIC, ε, γιατί αυτό σημαίνει ότι γίνεται ειδική μεταχείριση ορισμένων φορέων και κάποιες ε, λέξεις όπως ε, εμπορικός ή δημοσίως υποστηριζόμενοι φορείς δεν νομίζουμε ότι είναι οι κατάλληλοι. Ίσως θα ήταν καλύτερο να, το, να χρησιμοποιούνται άλλοι όροι. Όσον αφορά τώρα το θέμα που ετέθη για την UNESCO που μας πηγαίνει πίσω στο 2005 Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει για την επταετή περίοδο και το ίδιο θα ίσχυε και για τον περιορισμό στο πλαίσιο το, της οδηγίας για τα απτικοακουστικά. Υπάρχει ένα επιχείρημα για την αύξηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα και την ε, άσκηση πίεσης ε, προς τα πάνω στις διάφορες χώρες ε, που συμμετέχουν. Όσον αφορά τώρα την οικονομική διευκόλυνση, υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με το κατά πόσο μπορούν να ζητήσουν, να ζητήσουν οι τράπεζες κολάτερας εγγύησης. μπορούν να το κάνουν αυτό βεβαίως στο πλαίσιο συμπράξεων που ε, υποστηρίζονται. Μερικά ακόμα πράγματα θα ήθελα να πω. Ναι, ναι, Θέλουμε να κινηθούμε προς την απλοποίηση. Υπάρχουν ήδη μεταρρυθμίσεις ε, που σημαίνουν ότι είναι απλούστερα όλα αυτά και προσπαθούμε να τις συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και η χρήση των καταποκοπήν ποσών ε, είναι χρήσιμη, ειδικότερα στο πλαίσιο ε, της ψηφιοποίησης. 20.000 ε, είναι, είναι το flat rate, ενώ ε, για τις μεταφράσεις είναι διαφορετικό το επίπεδο ανάλογα με τον αριθμό των μεταφράσεων που λαμβάνουν χώρα. Συμφωνούμε και με την ύπαρξη περισσότερων ταινιών για τα παιδιά ε, και τα σχετικά φεστιβάλ, την προώθηση των παιδικών ταινιών. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα της παραγωγής ταινιών ε, που δυστυχώς ε, υπάρχει κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες και πολύ λιγότερο στις υπόλοιπες. Συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο. Σας ευχαριστούμε τα μάλα. Εγώ νιώθω κάποια αματέωση. Ελπίζω ότι κάποια από αυτά τα οποία έχουμε παρατηρήσει θα τα δεχτείτε πράγματι. Εντάξει, καλά είναι, καλές είναι Αλλά αυτό το είχε αναφέρει η κυρία Τρίπελ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω κυρία Ντασίλβα να μας πείτε και εγγράφω τι είναι αυτά με τα οποία δεν συμφωνείτε. Θα είναι χρήσιμο να μπορέσετε να αναφέρετε στους συναδέλφους, στην κυρία Κώστα και στους κοιόδης ποια είναι αυτά τα οποία θα τίνετε να απορρίψετε. Να έχουμε ένα κατάλογο λοιπόν γραπτό. Είναι πολύ δύσκολο να τα θυμηθώ όλα αυτά που είπατε. Δώστε μας λοιπόν αυτόν τον κατάλογο απορρίψεων θα είναι πιο εύκολο για την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές να λειτουργήσουν. Μπορώ να σας το ζητήσω αυτό ή είναι υπερβολικό. Εντάξει, πολύ ωραία. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν, δεν έχει νόημα τώρα η κυρία Κώστα να απαντήσει. Όχι. Σας παρακαλώ, έχουμε ακούσει ήδη. Ας ε, χωνέψουμε όλα αυτά τα στοιχεία, ας πάρουμε τα στοιχεία γραπτά από την Κομισιόν και τότε η Σίλβια μαζί με τους σκιώδεις συζητητές θα πρέπει να επανέλθει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται τώρα να το ε, επαναλάβουμε. Ναι, η Σίλβια. Καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Δύο μόνο πράγματα. Να πω στους συναδέλφους που πήραν το λόγο ότι με τα θέματα τα οποία έθεσαν δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί τους και πρέπει να τους το πω αυτό. Δεύτερον, θα μπορούσα ίσως να δώσω απαντήσεις στην Επιτροπή επί τη βάση των ε, αποφάσεων ή μάλλον των προτάσεων που θα μας κάνουν αλλά εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για τον πολιτισμό από αυτήν την οποία ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Σε ευχαριστώ πάντως ε, για την προσπάθεια την οποία έκανε. Σε ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έκανε κάποιες, ε, θα έλεγα, πρώτες νήξεις ε, των θέσεών της για το πρόγραμμα Creative Europe. Σας ευχαριστώ όλους. Οι συντονιστές έτσι και αλλιώς συναντήθηκαν χθες το απόγευμα. Ενημερωθήκατε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σήμερα το πρωί. Θα συναντηθούμε πάλι στις 18 Δεκεμβρίου. Καλή σας όρεξη.